Καλημέρα σας και χρόνια σας πολλά. Ξεκινάει η συνεδρίαση. Ο συνήθως θα ξεκινήσουμε από την ημερήσια διάταξη. Να αναφέρω πρώτα απ' όλα πως υπάρχουν αιτήματα αλλαγής Τη σημερινή διάταξη το αίτημα τη κυρία Ζαμπόρσκα η οποία είναι η αρμόδια για την, γνωμοδοτήσει πρωτοβουλία πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Συμβολή Ισότητα στην καταπολέμηση της νεανικής εγκληματικότητας. Θα συζητηθεί αλλά θα συζητηθεί μόνο σήμερα παρά το ότι αναβλήθηκε η ψηφοφορία. Η δε κυρία Γιανακουδάκη, η οποία είναι υπεύθυνη για την ε, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και την καταπολέμησή της και αυτή η ψηφοφορία θα αναβληθεί, αλλά πάλι το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη, οπότε θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Τώρα, Ο φάκελος για την ε, αποστολή στην Ισλανδία έχει φύγει από την ημερήσια διάταξη γιατί δεν μπορέσαμε να συντάξουμε την έκθεση. Συμφωνείτε με τις αλλαγές αυτές στην ημερήσια διάταξη. Ωραία, προχωράμε στο επόμενο σημείο το οποίο είναι οι ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Σημείο 4 έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης ε, της ε, Δευτέρας Σεπτεμβρίου. θα πρέπει να είναι τα πρακτικά μέσα στα εγγραφά σας. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση μέχρι το τέλος σημερινής συνεδρίας, θεωρούμε ότι τα πρακτικά εγκρίνονται. Οπότε... Περνάμε κατευθείαν στο σημείο υπαριθμών 5 δηλαδή η έκθεση της κυρίας Γιάννα Κουδάκη η γνωμοδότηση δηλαδή που αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Η αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Ελευθεριών. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Γιάννα Κουδάκη για να μας κάνει κάποιες ε, παρατηρήσεις και μετά θα μπορέσουμε να το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Ξέρετε πως ε, αυτό το συζητήσαμε ήδη στις 2 Σεπτεμβρίου. Να ε, σας πω πως η Επιτροπή Ελευθεριών εξήγαγε μία δημόσια κρόαση 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Γιανακουδάκη. Παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους. Ήρθα εδώ πέρα να σας μοιράσω τα μικρόβια μου καθοδόν προς την Ελλάδα. Είχαμε γύρω στις 100 τροπολογίες, οι οποίες κατά βάση λένε τα ίδια πράγματα. Οπότε τι προσπαθούμε να κάνουμε, να τις ενώσουμε και να βγάλουμε κάποιες συμβιβαστικές για να μην κάνουμε τα πράγματα δύσκολα. Φαίνεται πως όλοι συμφωνούμε. Το μόνο θέμα που δεν είναι καν επίμαχο. Είναι πως κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι ποινές φυλάκισης, δηλαδή αντί να πούμε πως θα ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές 5-6 χρόνια κτλ. Αυτό νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να ψηφιστεί. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα συγκεκριμένη ποινή για δύο λόγους, γιατί αν κάνω αυτό που θέλω θα προτείνω πολύ ψηλέ ποινέ, αλλά δεν νομίζω πως θα περάσει κιόλα και μπορεί και να εμποδίσει την γνωμοδότηση και δεν θέλω να κολλήσουμε σε λεπτομέρειες όταν έχουμε πιο σοβαρά πράγματα. Δεν ξέρω τώρα αν αυτά που λέω μεταφράζονται σωστά, ελπίζω να μεταφράζονται. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι το εάν θα πρέπει να μπλοκάρουμε ή να ε, αφαιρέσουμε κάποια πράγματα. Ε, είμαι και κρυωμένη, συγγνώμη. Υπάρχουν πάλι διαφορετικές απόψεις, αλλά νομίζω πως μπορούμε να, να τα συμπεριλάβουμε και τα δύο. Οπότε θα ήθελα να μάθω εάν εσείς θέλετε μία συνάντηση των συντονιστών ή να γίνει μέσω διαδικτύου. Χτες ψήφισε η Επιτροπή Προπολογισμού. Η Επιτροπή Πολιτισμού, με συγχωρείτε, η οποία το βλέπει ως ε, τεχνικό ζήτημα, δεν το κοιτάει από τη σκοπιά του φίλου ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε θα είναι δύσκολα τα, τα πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες, γιατί είναι πολύ καλές τροπολογίες και ενίσχυσαν την έκθεση. Οπότε τώρα αναμένω τα σχόλιά σας. Εντάξει, σας ευχαριστούμε κυρία Γιανακουδάκη. Σας ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα αυτή παρέμβαση. Ποιος θέλει το λόγο για σχόλια. Κανείς. Α, όχι. Η κυρία Ζαμπόρσκα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και την κυρία Γιανακουδάκη για την εξαιρετική της εργασία. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μπορέσαμε να δούμε τα πράγματα όπως είναι, όπου το δείχνουν αυτό και οι τροπολογίες. Ξέρω ότι πρόσφατα εγκρίθηκε ανακοίνωση με παρόμοιο θέμα που μιλούσε για την ελευθερία του λόγου στο δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ Αυτόν που λέει η Κομισιόν και αυτόν που έχει πετύχει η, επιτοχή, η Επιτροπή μας. Το ΕΛΚ στηρίζει την έκθεση. Ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόρκα τώρα. Ο κύριος Σοβέν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επί του κειμένου θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το κείμενο αυτό Με απασχολεί ένα ζήτημα και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής όλους. Το κείμενο της Κομισιό μιλάει για τα παιδιά. Και μιλάμε για ένα άτομο το οποίο δεν έχει φτάσει στην σεξουαλική οριμότητα. Στο κείμενο της Επιτροπής μιλάμε για κάτω από τα 18 χρόνια μιλάμε για την σεξουαλική ενηλικίωση και άλλες φορές γίνεται λόγος για κάτω από 18 χρόνια. Δηλαδή σε άλλα σημεία μιλάμε για σεξουαλική ενηλικίωση και σε άλλα σημεία για κάτω από τα 18 χρόνια. Ποια είναι η σωστή η πρόταση, ποια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, θα πρέπει να μιλήσουμε για σεξουαλική ενηλικίωση ή για κάτω από τα 18. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στην κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πως ήθελε να απαντήσει η κυρία Γιανακουδάκη, αλλά ίσως καλύτερα να απαντήσει μια και καλή στο τέλος. Πράγματι πρέπει να γίνει η διάκριση τι εννοούμε σεξουαλική ενηλικίωση και 18 έτη. Βεβαίως η παιδική πορνογραφία ανεξαρτήτως ηλικίας είναι αδίκημα. Αλλά γενικά νομίζω καλό είναι να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό. Δεν είναι θέμα γυναικείο τόσο. Αφορά τους νέους αλλά και τα δύο φύλλα. Και δυστυχώς αφορά και τα δύο φύλλα και τους, ε, όσον αφορά και τους δράστες. Δηλαδή μπορεί να είναι και γυναίκες. Να πω πως έκανα μία παρατήρηση για τα προγράμματα θεραπείας. Πρέπει να δούμε πως ε, θα πρέπει να διαγραφεί από το ίντερνετ ότι είναι τέτοιο και όχι μόνο να σβηστεί, αλλά βεβαίως να δούμε τι θα κάνουμε και με τη θεραπεία των δραστών και με την ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Νομίζω υπάρχει στην Αγγλία εκεί πέρα μια γραμμή βοήθειας όπου μπορεί να τηλεφωνήσει κανείς πριν γίνει δράστης. Και μπορούμε ίσως να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να εμποδίσουμε τα δικήματα σε αυτό το τομέα. Γιατί οτιδήποτε συμβαίνει εδώ πέρα είναι ήδη δηλαδή αρκετά άσχημο για τα παιδιά τα οποία αφορά. Ευχαριστώ κυρία Μπάουρ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Μαρίνα για τη γνωμοδότηση αυτή. Να κάνω δύο σύντομες παρατηρήσεις. Όσον αφορά το όριο ηλικία, όταν μιλάμε για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν υπάρχει αμφιβολία πως το όριο θα πρέπει να είναι 18 χρόνια όχι λιγότερο. Υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια να αναγνωρίζουμε σε όλες τις περιπτώσεις όπου μιλάμε για παιδιά πως το όριο ηλικίας είναι τα 18 χρόνια. Είτε μιλάμε για σωματεμπορία, είτε μιλάμε για τα δικαιώματα των παιδιών, είναι σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ 18 χρόνια. Το δεύτερο ζήτημα, όπως ανέφερε και η Μαρίνα, είναι αυτό το να αφαιρούμε ή να μπλοκάρουμε τα site. Από τη σκοπιά της τεχνολογίας πιθανότατα η προτεραιότητα είναι να, να σβηστούν, να, τα, να αφαιρεθούν. Πιθανώς υπάρχουν και άλλες συμπληρωματικές πηγές για να μπουν αυτά τα υλικά ε, και ίσως να είναι ίσως πιο προβληματικό το ζήτημα και ίσως η τεχνικοί που ασχολούνται εκεί με το ίντερνετ είναι υπέρ του μπλοκαρίσματος, όχι της αφαίρεσης, του κατεβάσματος. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να ζητήσουμε στενότερη συνεργασία. Δεν ξέρω, κάποιον απεσταλμένο στη ΣΥΠΑ έχουμε για την προστασία των δεδομένων. Ίσως σε αυτή την περίπτωση το άτομο αυτό να έχει και κάποια ευθύνη για να σβήνει αυτές τις σελίδες που φιλοξενούνται στις ΙΠΑ γιατί πολλές από αυτές τις σελίδες είναι είτε στη Ρωσία είτε στην Αμερική ευχαριστώ ευχαριστώ κυρία Μπάουερ θα δώσω τον λόγο στην κυρία Μποσκούρτ ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε καταρχήν ευχαριστώ την εισηγήτρια. Έχω κάποιες ερωτήσεις γιατί είπε η εισηγήτρια πως θα προσπαθήσει να δει το ζήτημα του να μπλοκάρουμε <clears throat> ή να απομακρύνουμε να το βάλει σε έναν συμβασμό. Για μένα δεν είναι αυτή η σημαντικότερη συζήτηση. Μας έχει να το λύσουμε. Βέβαια είμαι περίεργη για το πώς θα το λύσουμε. Δεύτερο, Έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες, αλλά έχω και κάποιες ε, τροπολογίες, αλλά το ερώτημα είναι πράγματι το όριο ε, ε το οποίο συχνά ε, φαίνεται πως αποτελεί εμπόδιο για την δίωξη αυτών των ανθρώπων. Και έτσι μπορούν να ξεφεύγουν από τη δίωξη. Κάτι άλλο. τη στιγμή που γίνεται σε ένα θεσμικό πλαίσιο η κακοποίηση, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι σε έναν υπηαγωγείο ας πούμε ή κάτι τέτοιο, ε, δηλαδή εκεί όπου κανείς εμπιστεύεται τα παιδιά του ότι είναι σε καλά χέρια, να αποτελεί αυτό κάτι το επιβαρυντικό για την ε, πίνη να καθιστά δηλαδή το αδίκημα σοβαρότερο. Ευχαριστούμε κυρία Μποσκούρτ, πράγματι είναι σοβαρό το πρόβλημα αυτό. Κύριε Κοντάκη, βλέπω πως, θέλ, πως θέλετε να απαντήσετε και να κάνετε κάποια τελικά σχόλια. Right, Καταρχήν, σε σχέση με το θέμα του παιδιού, πώς ορίζεται. Κάνουμε μία διάκριση, διότι αυτό ήταν ένα πρόβλημα με την πρόταση της Κομισιόν. Μία από τις τροπολογίες λέει ότι έχουμε ε, παιδιά, μιλάμε για παιδιά τη στιγμή που βρίσκονται υπό κυδαιμονία. Νομίζω 16 είναι στο Ενωμένο Βασίλειο, στο Βατικανό 12. Άρα ε, μπορούμε να μιλάμε για παιδί και ε, έναν έφηβο ο οποίος είναι μέχρι τα 18. Αν και υπάρχει σεξουαλικό έγκλημα και στις δύο κατηγορίες, μπορούμε να μιλήσουμε για συνένεση, για ηλικία συνένεσης που είναι τα 17. Αν κάποιος βεβαίως υποχρεωθεί ή υποστεί σεξουαλικές σχέσεις, τότε υπάρχει μια διαφοροποίηση. Μιλάμε λοιπόν για παιδιά και, και εφήβους ναι, μιλάμε και για τα δύο φύλλα. Όταν μιλάμε για βία, για σεξουαλική ε, ε, βία και μπορούμε να πούμε ότι οι θύτες ε, προέρχονται και από τα δύο φύλλα, γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε ομάδες ανδρών και γυναικών, δηλαδή άνδρες και γυναίκες, σύζυγοι γιατί το κάνουν οι γυναίκες, ίσως γιατί υφίστανται πίεση από τους συζύγους. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε γιατί η γυναίκα παίζει το ρόλο του, ε, του δευτέρου βιολιού, αν μπορώ να το πω έτσι. Βεβαίως υπάρχουν ε, συμβούλια, δηλαδή ε, παροχή συμβουλών για τα δύο φύλλα. Υπάρχει ένας αριθμός ελεύθερης κλίσης και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και να παρέχονται ε, συμβουλές και προς την οικογένεια των θητών γιατί συναντήθηκα με ορισμένες από αυτές τις οικογένειες και είναι πολύ ε, δύσκολο όταν πιστεύεις ότι έχεις παντρευτεί έναν καλό οικογενειάρχη και κάποια στιγμή συλλαμβάνεται γιατί ήταν ένας θήτης και καταλαβαίνετε ότι αυτό πλήττει ολόκληρη την οικογένεια. Γι' αυτό χρειάζεται βοήθεια και, της, και η οικογένεια. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε έναν ιδεώδη κόσμο θα ήταν σκόπιμο να διαγράψουμε αυτό το σκέλος του διαδικτύου. Εάν λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να το διαγράψουμε, άρα το αφήνουμε. Τα παιδιά, οι, οι έφηβοι, οι ενήλικοι ξέρουν ότι έχουν ανεβάσει τις ε, φωτογραφίες τους στο ίντερνετ, άρα ξέρουν ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο βίας. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει αυτό το μπλοκάρισμα αλλά βεβαίως η διαγραφή είναι βεβαίως προτεραιότητα. Ξέχασα το τελευταίο σημείο. Η κυρία Μπάουερ, όχι με συγχωρεί, η κυρία Μποσκούρτ είπε για πόσο χρονικό διάστημα θεωρείται η αδικοπραξία αδικοπραξία. Εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Εμείς έχουμε περιπτώσεις όπου τα παιδιά ε, ε, αποτέλεσαν θύμα βίας και ήταν πολύ, σε πολύ μικρή ηλικία. Δεν νομίζω θα πρέπει να αλλάξει το δίκαιο στις χώρες, το, το ποινικό δηλαδή θα πρέπει να προβούμε σε συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω κατά πόσο από, από τεχνικής ή ουσιαστικής πλευράς μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω ότι απάντησα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει και μία Συμπληρωματική ερώτηση. Θα ήθελα να επιμείνω εκ νέου σε αυτό το πρόβλημα. Άρθρο 2 της πρότασης της Επιτροπής. Άρθρο 2α. Ορίζει το παιδί ως ένα πρόσωπο κάτω των 18. Κάτω των 18. Άρα όλα, ό,τι ισχύσει θα ισχύσει για τα παιδιά κάτω των 18. Όμως στο άρθρο 3 στο, στα σημεία 2 και 3 η Επιτροπή αναφέρει, μιλάει για ένα παιδί το οποίο δεν έχει φτάσει στη σεξουαλική οριμότητα. Για τη Γαλλία είναι τα 16 χρόνια, δηλαδή το άρθρο 2 μιλά για όλα τα παιδιά κάτω των 18 και το άρθρο 3 λέει ναι αλλά μόνο για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν φτάσει στη σεξουαλική οριμότητα. Δηλαδή, στη Γαλλία είναι τα 16 χρόνια. Όταν διαβάζω λοιπόν ε, το άρθρο 2, τα άρθρα 2 και 3, βλέπουμε ότι μεταξύ 16 και 18 δεν υπάρχει εφαρμογή του νόμου. Άρα θα πρέπει να μιλάμε για τα 18 χρόνια και όχι για σεξουαλική οριμότητα. Νομίζω ότι καμία τροπολογία δεν έχει υποβληθεί επί του θέματος. Εγώ οφείλω να ομολογίζω ότι αυτές, οι δύο προτάσεις αυτές δύο προτάσεις δεν τις είχα εξετάσει, μου είχαν διαφύγει. Αν λοιπόν συμφωνήσουμε όλοι για τα 18 χρόνια και όχι τη σεξουαλική οριμότητα, τότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να υποβάλουμε μια προφορική τροπολογία. Ήμουν σαφής, τι θα κάνουμε δηλαδή μεταξύ τα 16 και 18. Θα πρέπει να εμείνουμε στα 18 χρόνια και να μην μιλάμε για σεξουαλική οριμότητα. Η κυρία Γιανακουδάκη, από όσο κατανοώ, 18 είναι η, η, σωστή ηλικία. Απλώς κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ παιδιών και εφήβων, αλλά η ουσία αφορά τα 18 χρόνια. Εάν θεωρείτε ότι το ζήτημα θα πρέπει να γίνει σαφέστερο, τότε θα πρέπει να, να καταστεί σαφέστερο μέσω προφορικής Μία προφορική τροπολογία. Ναι, πράγματι, πιστεύω ότι στο άρθρο 3, σημεία 2 και 3, θα πρέπει να μην γίνεται λόγος για σεξουαλική οριμότητα. Αλλιώ δεν, δεν γίνεται κατανοητό το κείμενο και είναι και λίγο αντιφατικό. Δεν καλύπτει όλο το ηλικιακό φάσμα. Η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή μας της 29 και 30 Νοεμβρίου και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα ψηφίσει στα μέσα Μαρτίου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γιανακουδάκη και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση Ζαμπόρσκα που αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας για, για την ισότητα ανδρών και γυναικών στην καταπολέμηση εγκληματικότητας των νέων. Ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε μία συνάντηση με εμπειρογνώμονες τον Ιούνιο και στις 28 Σεπτεμβρίου είχαμε μία συζήτηση. Είχαμε 150 προτινόμενες τροπολογίες και σήμερα άλλη μια δυνατότητα, ακόμα μια δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ζαμπόρσκα που θα μας κάνει ορισμένα εισαγωγικά σχόλια. Έχετε το λόγο κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την συνεργασία και για την προσπάθεια να βελτιωθεί το σχέδιο έκθεσης. Θεωρώ πως όλοι μας, τα μέλη εδώ της Επιτροπής Γυναικών, ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για την καταπολέμηση της μάστιγας αυτής της κοινωνίας. Δηλαδή της εγκληματικότητας των νέων. Όπως είπατε, κυρία Πρόεδρε, έχουμε λάβει και 147 τροπολογίες και επειδή χρειάζεται χρόνος για τη μετάφραση, υπέβαλα εγώ το αίτημά μου περί αναβολής της ε, ψηφοφορίας και ευχαριστώ την Πρόεδρο και τους συντονιστές που το δέχτηκαν σήμερα θα συζητήσουμε τροπολογίες και μετά, όπως είπε η κυρία Γιανακουδάκη, θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια συμβιβαστική πρόταση να συναντηθούμε με τους κοιόδης συγητές. Να πω κάτι για τις τροπολογίες, οι μισές περίπου αφορούν παραπομπές, έγγραφα, γεγονότα και οι υπόλοιπε είναι συστάσεις ή αιτήματα προς την Κομισιόν ή τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση. Οι τροπολογίες αυτές αναφέρουν το ότι έχουμε πολλά να κάνουμε για να διασφαλιστεί η καλύτερη ισότητα ανδρών και γυναικών στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων παρά το ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το θέμα δεν είναι έλλειψη νομοθεσίας αλλά η εφαρμογή της νομοθεσίας. Προσπάθησα λοιπόν να μειώσω και τον αριθμό των τροπολογιών και κατέληξα σε 11 συμβαστικές τροπολογίες. Αναθέμα και τι επόμενες μέρες θα έρθω σε επαφή με του συναδέλφου και θα του πληροφορήσω για το ποιες ε, θα ήθελα να γίνουν συμβαστικέ. Να σταθώ τώρα σε κάποιες συγκεκριμένες τροπολογίες. Θα μιλήσω γενικά, όχι για συγκεκριμένες. Υπάρχει π.χ. μια τροπολογία Υπήρχε μία που αναφέρεται στη μια γενική, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η τροπολογία επεκτείνει ακριβώ αυτόν τον ορισμό με βάση την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Παρά το ότι σε συζητήματα ουσία σκεπτικό είναι καλό, δεν νομίζω πως μπορούμε να αλλάξουμε έναν ορισμό που υπάρχει σε ένα άλλο γενικά γνωστό έγγραφο και επειδή συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει η Μέρη Χάνιμπαλ εγώ έμεινα μόνο στη μητρότητα και στο δικαίωμα των γονιών να διαλέγουν την απασχόλησή τους οπότε δεν έχω συμπεριλάβει τον ορισμό της οικογένειας για να συμπεριλάβω τις διάφορες μορφές συγκατοίκησης που υπάρχουν στη σημερινή κοινωνία. Υπάρχει μετά μια τροπολογία που αναφέρεται σε διαφορετικές απειλές τις οποίες εκτίθενται τα παιδιά όταν ζουν στη φτώχεια. Υποστηρίζω πλήρως αυτή την τροπολογία, αλλά για να αποφευθούν παρεξηγήσεις πρέπει να μιλήσουμε για ακραία φτώχεια. Γιατί φέτος είναι το έτος καταπολέμησης της έσχα της ένδυας. Και θα πρέπει να μπορέσουμε να αποδεχτούμε μια τέτοια προφορική τροπολογία. Κύριο Σιμάνσκι άλλαξε λίγο τη διατύπωση αλλά νομίζω πως αυτό το οποίο προτείνει και αυτό το οποίο έχω στο αρχικό σχέδιο ε, είναι δύο πράγματα συμβατά. για να μπορέσουν να εκφράσουν τις φιλοδοξίες τους οι νέοι. Να μιλάμε λαμβάνω μόνο το τι γίνεται τώρα με τους νέους. Θα βρούμε λοιπόν μια συμβιβαστική λύση νομίζω. Μια... Σε μια άλλη τροπολογία μιλάμε για διάφορες μητρικές γονικές άδειες ε, και πρέπει νομίζω να φέρουμε και την άδεια υιοθεσία. Νομίζω σωστό είναι να μπει εδώ πέρα. Υπάρχουν οι 70, οι 71, 77, 78, 85, 139, 146 από τρεις συναδέλφους Αυτές οι δέκα τροπολογίες έχουν κάτι κοινό. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι θέλουν από τις σχετικές παραγράφους να αφήγει η εξάσκηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των γονέων. Έχω μια ερώτηση. Δεν νομίζω πως είναι εδώ κάποιος από τους συναδέλφους, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί επιμένουν σε σχέση με την εγκληματικότητα των νέων να μιλάμε για την ευθύνη των γονιών. Εξπακούεται πως η ανατροφή των παιδιών ε, δεν είναι εγγύηση για το μέλλον αυτών των νέων αλλά σε αρκετές χώρες οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των παιδιών τους μέχρι αυτά να φτάσουν μια ηλικία. Εάν θέλουν ε, να συμπεριφέρονται υπεύθυνα γονείς πρέπει να δούμε και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Υπάρχει σχέση μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των γονιών και της καταπολέμησης εγκληματικότητας των νέων. Σκοπεύω να μιλήσω με τους τρεις αυτούς συναδέλφους. Γιατί θέλουν να αφαιρεθούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των στην προηγούμενη θητεία. Η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια έκθεση της κυρίας Μπατζελή των σοσιαλιστών που έκανε λόγο για τον ρόλο της κοινωνίας, οικογένειας ε, και γυναίκας στην καταπολέμηση της ε, νεανικής εγκληματικότητας. Νομίζω λοιπόν πως εκεί πέρα υπήρχε μια συνένεση στο ότι η οικογένεια έχει να παίξει ένα ρόλο κλειδί στην καταπολέμηση της νεανικής εγκληματικότητας. Και ακόμη μια τροπολογία όπου Αναφέρομαι σε αρκετές οργανώσεις, εταιρείες, κοινότητες που θα πρέπει να εμπλακούν στην καταπολέμηση της νεανικής εγκληματικότητας. Το αναφέραμε αυτό κατά τη διάρκεια και των προηγούμενων και το, της ακρόασης. Υπάρχει μια τροπολογία που λέει πως ο κατάλογος αυτός ε, των οργανώσεων δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες και καταλαβαίνω γιατί. Η ζωή δείχνει πως οι θρησκευτικές κοινότητες εμπλέκονται σε μέρη και σε κοινότητες που ε, είναι υψηλού κινδύνου όσον αφορά την εγκληματικότητα και επιτυχώς. Εγώ έχω λάβει μέρος σε πολλές συζητήσεις π.χ. για τους Ρώμα στη Γαλλία και προέκυψε πως ε, κράτη όπου υπάρχουν μεγάλες κοινότητες Ρωμά οι δραστηριότητες εκκλησιών ε, που είναι κάτι το οποίο επενείται. Δεν νομίζω πως ε, θα χαλάσει η έκθεση αν μείνει αυτή η αναφορά εάν αφαιρθούμε στο ρόλο της οικογένειας, των σχολείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, δεν θα γίνει και τίποτα άμα μείνουμε σε και οι εκκλησίες Επίσης, γιατί θέλετε να σταματήσει η πολιτική της μηδενικής ανοχής έναντι ενηλίκων που ε, παρακινούν τα παιδιά να κάνουν κάποιο έγκλημα. Ε, καμιά φορά είναι οι γονείς που το κάνουν αυτό. Καμιά φορά επειδή τα παιδιά δεν είναι νομικά, ποινικά υπεύθυνα, τα βάζουν οι γονείς να κάνουν αυτά τα αδικήματα. Ε, όχι, πρέπει να μην διαπηδείξουμε καμία ανοχή στους γονείς αυτών των παιδιών που αλλάζουν έτσι τη ζωή των παιδιών τους. Θεωρώ πως την έκθεσή μου καλό θα ήταν να πούμε πως το κόστος της ισορροπίας της ε, δουλειάς και της οικογένειας θα πρέπει να το επομίζεται το κράτος. Γιατί το κράτος πρέπει να φροντίσει πως η πολιτική της μη διακριτικής μεταχείρισης, η δημογραφική πολιτική και η ισορροπία ζωής και εργασίας θα πρέπει να υπάρχουν. Οπότε το κράτος θα πρέπει να λάβει αυτό το κόστος. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για την αδιαμητρότητα, για την προστασία των εργαζομένων γυναικών και είχαμε κάποιες επιφυλάξεις γιατί λέγανε πως το κόστος ε, αυτό το επομίζονται οι εργοδότες οπότε δεν ήθελαν η άδεια να επεκταθεί ή να λαμβάνουν οι γυναίκες το 100% του μισθού. Η δημογραφική πολιτική νομίζω είναι προς το συμφέρον του κράτους και το κράτος θα πρέπει να χρηματοδοτεί ε, αυτή την πολιτική. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια κίνηση για να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Επίσης, αναφέρθηκαν κάποιοι όροι για το πώς ζουν οι νέοι στα σοφρονιστικά καταστήματα και κάποιοι είπαν πως θα πρέπει να μπορούν να εξασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. π.χ. να μπορούν να προσεύχονται στο, κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Δεν είμαι πάρα πολύ υπέρ, όχι γιατί είμαι κατά των μουσουλμάνων, απλά γιατί στη φυλακή και στα σοφρονιστικά α, καταστήματα δεν υπάρχουν μόνο μουσουλμάνοι, πρέπει να αφαίρουμε και τα άλλα δόγματα άμα είναι έτσι. Γιατί έτσι φαίνεται πως μόνο μουσουλμάνοι είναι οι κρατούμενοι. Αυτό είναι διακριτική μεταχείριση. Δεν είναι σωστό. Ε, δεν πρέπει να δημιουργείται τέτοια εντύπωση. Πρόθεσή μου είναι για τις ε, τροπολογίες. Να σας πω πως συμφωνώ με τη συντριπτική του πλειοψηφία ανεξαρτήτως ε, του ποια ομάδα της υπέβαλε. Βλέπω εδώ πέρα πως υπάρχει μια πραγματική επιθυμία να βελτιωθεί η διατύπωση για την καταπολέμηση της νεανικής εγκληματικότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Ζαμπόρσκα, που μας εξηγήσατε τις τροπολογίες. Και τώρα η κυρία Τόμσεν. Ευχαριστώ. Δυστυχώς λείπει η συγγήτριά μας και γι' αυτό δεν μπορεί να μας εξηγήσει η ίδια τις τροπολογίες, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να σχολιάσω ορισμένα από αυτά που είπατε. Δεν θα διαχωρίσω καλές από κακές επιρροές αλλά θα ήθελα να πω ότι διαφέρει η κατάσταση από χώρα σε χώρα στις σκανδιναβικές χώρες τουλάχιστον θα θεωρούνταν πολύ αρνητικό να παίξει κοινωνικό ρόλο η Εκκλησία. Πληρώνουμε 15% των μισθών μας. 50. 50% των μισθών μας για το κράτος. I'm not saying what one is better or worse or uh, uh, putting a value on that. Και επομένως δεν σχολιάζω εδώ, δεν κρίνω, αλλά λέω ότι είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι τα ίδια τα πράγματα σε όλες τις χώρες και για μας δεν έχει νόημα να μιλάμε για κοινωνικό ρόλο της Εκκλησίας είτε πρόκειται για τους Ρωμά είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Είναι το κράτος που πρέπει να κάνει τη δουλειά αυτή. Ευχαριστούμε κυρία Τόμσεν. Ο κύριος Σοβέν. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήθελα η Επιτροπή μας να γίνει χώρος ε, υπέρ κατά της Εκκλησίας το θέμα της νεανικής εγκληματικότητας είναι πολύπλοκο και κανείς δεν μπορεί να πει ότι μόνο το κράτος μπορεί να το λύσει. Αν τα κράτη είχαν τη δυνατότητα και την εξυπνάδα να το λύσουν, δεν θα χρειαζόταν και εμείς να το συζητάμε. Ξέρουμε ότι τα κράτη πρέπει να βασιστούν, να στηριχθούν σε ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό για να αντιμετωπίσουν την νεανική εγκληματικότητα. να χορηγηθεί βοήθεια για τα παιδιά, στα παιδιά που έχουν αφαιθεί μόνα τους, που είναι εγκαταλελειμμένα στους δρόμους και ξέρουμε ότι γενικά οι εκκλησίες, όχι μία εκκλησία, έχουν έναν κοινωνικό ρόλο να παίξουν, όπως και οι αγνωστικιστικές οργανώσεις εξάλλου. Μιλάμε για κοινωνικό ιστό γενικότερα που μπορεί να παίξει το ρόλο του είτε πρόκειται για θρησκευτικού χαρακτήρα οργανώσεις χωρίς να λέμε ότι είναι μια εκκλησία προτιμότερη από την άλλη αυτό είναι μια πραγματικότητα και θα ήταν κρίμα να δηλώσουμε εκ των προτέρων ότι δεν θέλουμε τους μεν και δεν θέλουμε τους δεν να παίξουν κανένα ρόλο. Όπως ξέρετε στη Γαλλική Δημοκρατία ο χαρακτήρας του κράτους είναι κοσμικός αλλά παρόλα αυτά στηρίζεται σε όλους αυτούς τους παράγοντες, θρησκευτικούς και μη. Ευχαριστούμε. Σιμάνσκι. ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κανένας αντικληρικαλισμός εδώ. Ίσως πρόκειται για παρεξήγηση δεν είναι θέμα ούτε τιμής ούτε ταπεινότητος αλλά νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε τη βοήθεια οποιασδήποτε ομάδας μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα. Και στις πλουσιότερες χώρες μέλη δεν μπορεί το κράτος να τα λύσει όλα. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι τομείς της ζωής όπου το κράτος δεν μπορεί να κάνει τίποτα και χρειάζονται θελοντές και εθελόντριες. ανεξαρτήτως του κράτους. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το προσέξουμε γιατί δεν θέλουμε να φανεί ότι είμαστε επιτροπή που εξετάζει τα πράγματα είτε από θρησκευτική είτε από αντιθρησκευτική προοπτική. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις όχι συναισθηματικά. Πολλοί οργανισμοί στην Πολωνία ακόμη και φυλακισμένων οργανώσεις και φυλακές δεν έχουν αρκετούς πόρους και η ανέχεια αυξάνεται. Εδώ στην Ευρώπη σε πολλές χώρες μέλη και στη Δυτική Ευρώπη ακόμα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Κατανοώ λοιπόν τις προθέσεις όλων αλλά να μην υπάρξουν εδώ παρεξηγήσεις γιατί πιστεύω ότι δεν χρειάζεται συναισθηματισμός που θα μπορούσε να βλάψει το στόχο μας. Ναι. Ε, ευχαριστούμε η κυρία Φιγκερέντου. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Ε, ε, ήθελα να πω ότι η σκιώδης εισηγήτρια δεν βρίσκεται εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να παρέμβω λαμβάνοντας σε υπόψη αυτά που άκουσα και ε, με βάση τα όσα γνωρίζω. Θα ήθελα να πω ότι στη χώρα μου θα ήθελα να πω ότι τη βασική ευθύνη φέρει το κράτος και οι οικογένειες. Ε, ζούμε σε ένα κοσμικό κράτος. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη την συνεισφορά πολλών οργανώσεων και εκκλησιαστικών οργανώσεων και στη χώρα μου είναι πολύ μεγάλη αυτή η συμμετοχή και εδώ πρόκειται για μία παράδοση, προαιώνια παράδοση, διότι το κράτος στο παρελθόν δεν αναλάμβανε τέτοιες ευθύνες. Μετά από την 25η Απριλίου του 1974 ανέλαβε τις ευθύνες του το κράτος. 75. Και... Αλλά είναι γεγονός ότι σήμερα δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις διότι δυστυχώς η πολιτική λιτότητας οδηγεί σε σοβαρές ε, παλινοδίες και η ίδια η Καθολική Εκκλησία διαμαρτύρεται διότι η φτώχεια έχει τέτοια ευρύτητα πλέον και τέτοιες διαστάσεις που και η ίδια δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί. Συμμετέχουν και πολλές άλλες οργανώσεις. Επειδή προβάλλουμε μία πολιτική συζήτηση, εδώ θα πρέπει να μας απασχολήσει η κυβερνητική πολιτική, δηλαδή η συμμετοχή του κράτους στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων. Η φτώχεια και οι μεγάλες ανισότητες είναι τα αίτια της εγκληματικότητας των νέων Γι' αυτό το κράτος θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Πριν από την Επανάσταση εμείς γνωρίσαμε μεγάλη φτώχεια γιατί το κράτος δεν παρενέβαινε και η Εκκλησία δεν μπορούσε να δώσει φυσικά μία σοβαρή απάντηση. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ολοκληρωτικά το θέμα ολοκληρωμένα. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται μια κυβερνητική καθαρά πολιτική για να αντιμετωπίσει θέματα φτώχειας, ανισότητας και έτσι μόνο θα ε, καταφέρουμε να πατάξουμε την εγκληματικότητα. Δεν έχει σημασία να μιλήσουμε, να δώσουμε δηλαδή μία άλλη εικόνα σε σχέση με τη συμμετοχή της Εκκλησίας. Εν πάση περιπτώσει, είτε είναι ε, θρησκευτικές είτε κοσμικές οι παρεμβάσεις, σημασία έχει να καταπολεμηθούν τα αίτια της κακοδαιμονίας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Φιγκέιρεδο, η κυρία Σίνκλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ ε, βεβαίως όταν μιλάμε για θρησκεία υπάρχει μια συναισθηματική χρειά στη συζήτηση. Αν δείτε όλες τις επιτυχείς ε, ε, κοινωνίες, τις κοινωνίες που έχουν επιτύχει, βλέπετε ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ εκκλησίας και κράτους. Δεν είναι σωστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει σε ε, οποιαδήποτε ε, συμμετοχή, να επιβάλλει μάλλον σε θρησκευτικά σχήματα να συνεισφέρουν και να συμβάλλουν. Αλλά νομίζω ότι μιλάμε για μια εταιρική σχέση, για συμμετοχή του κράτους πρωτίστως, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείτε να επιβάλλετε στη θρησκεία τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να έχουμε μία ε, κάταντη δικτατορία την οποία να επιβάλλουμε είτε στο κράτος είτε στη θρησκεία. Η κυρία Τόμσεν, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν επιτέθηκα στην Εκκλησία. Απλώ θεωρώ ότι δεν ε, μπορούμε να επιβάλλουμε ένα μοντέλο. Κανένα δεν είναι καλύτερο από το άλλο. Απλώς ο ρόλος της Εκκλησίας είναι διαφορετικός από μια χώρα στην άλλη. Γνωρίζω ότι ιστορικά η Καθολική Εκκλησία έχει συνεισφέρει και έχει γίνει μεγάλη κοινωνική εργασία, αλλά αυτό δεν ισχύει στις χώρες όπου επικρατεί ο προτεσταντισμός, όπου η Εκκλησία διαδραματίζει διαφορετικό ρόλο. Είναι πιο περιορισμένη οι διακρίσεις οδηγούν στην εγκληματικότητα των νέων, ιδιαίτερα ως προς τους νέους μουσουλμάνους στις χώρες μας, επειδή δηλαδή δεν ενσωματώνονται στην κοινωνία, γι' αυτό επαναστατούν, γίνονται εγκληματίες. Και γι' αυτό στρέφονται στο τζαμί και στο τζαμί βεβαίως ε, μπορούν να γίνουν ακόμα, να μετατραπούν σε ακόμα πιο εχθρικά στοιχεία με βάση τη θρησκεία επειδή αποτελούν αντικείμενο ε, διάκρισης. Γι' αυτό με απασχολεί και αυτή η διάσταση του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τόμσεν και κυρία Παλανόβα. Ευχαριστώ. Και η δική μας ε, σκιώθης δεν είναι εδώ, αλλά συμμερίζομαι τις απόψεις αυτές από πλευράς φιλελευθέρων, διότι όλα αυτά συζητήθηκαν και οι, εμείς οι φιλελεύθεροι θεωρούμε ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε το ρόλο της Εκκλησίας και ε, τη συμμετοχή του κοσμικού κράτους. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για το ρόλο της κοινωνίας, της οικογένειας, της ατομικής οριμότητας και να μιλήσουμε και για μειονότητες ή νέους από ομάδες υψηλού κινδύνου και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα συνολικά σε σχέση με την κρίση, τη φτώχεια, την, ε, το δημογραφικό και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες και να μιλήσουμε υπέρ κατά της Εκκλησίας, γιατί αυτό δεν βοηθά. Στην πολιτική μας ομάδα δεν έχουμε εκπροσώπους από χώρες που την χάνουν υποστήριξη της Εκκλησίας. Επειδή είμαστε φιλελεύθεροι λοιπόν και εξαιτία αυτού έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση, αλλά δεν θέλουμε να πέσουμε σε μία αντίφαση εδώ. Ε, πρόκειται για μία νέα και δύσκολη έκθεση και δεν θα πρέπει να εκτεθούμε, να μην διαφωνήσουμε, να είναι χρήσιμη λοιπόν, να σταθεί χρήσιμη αυτή η πρόταση ψηφίσματος για τα κράτη-μέλη. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Ladies και κύριοι, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε με μια μικρή καθυστέρηση, γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε πια με τη συνεδρίασή μας. Χαίρομαι που έχω αναλάβει την Προεδρία, είναι έκπληξη. Βέβαια κάποιος από τους συναδέρφους είπε «Α, επιτέλους». Γιατί, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθώ να είμαι πρόεδρος στην Επιτροπή αυτή περιβάλλοντος. Επευκαιρία σας λέω ότι έχω παραιτηθεί πια από αυτή την επιθυμία, αλλά εν πάση περιπτώσει χαίρομαι που βασικές ιδέες. Καταρχήν, οι πρώτες σελίδες συμπεριλαμβάνουν το σχέδιο γνωμοδότησης, υπάρχει και η αιτιολογική σκέψη και στο τέλος συστάσεις. Και βεβαίως υπήρχε ένας περιορισμένος αριθμός σελίδων. Ήμασταν υποχρεωμένοι για κάτι τέτοιο. Το κείμενο βεβαίως μπορεί να τροποποιηθεί για να λάβει μία ε, πλέον πολιτική χρειά. Στις 10 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία υποβολής. 30 ε, Νοεμβρίου θα ψηφιστεί εδώ και το Μάρτιο του 2011 θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια, δηλαδή θα πρέπει να ψηφίσουν οι δύο επιτροπές, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δικαιωμάτων των Γυναικών. Εγώ θα λάβω υπόψη τα σχόλιά σας και θα τα διαβιβάσω στην κυρία Κιγιό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Ταραμπέλα. Αρχίζει η συζήτηση τώρα. Κυρία Παραφενόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο σκιώδης μας για αυτό το θέμα, η σκιώδης μας είναι η Σόφη Ιντβελτ που δεν παρίσταται και θα την αντικαταστήσω εγώ εφόσον είμαι και εγώ σκιώδης για την περίφ για το ίδιο θέμα. Βασιστήκαμε στην σχετική δήλωση της Κομισιόν από πέρι, την περσινή, που είχε προβλεφθεί να εξεταστεί από το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο, μετά αναβλήθηκε για το Φεβρουάριο και τώρα ξανααναβλήθηκε γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτών των ανισοτήτων στον υγειονομικό τομέα. Αν θέλουμε να βάλουμε το θέμα των φύλων εδώ θα χρειαστούμε σοβαρές τροπολογίες γιατί από άλλες εκθέσεις στην Επιτροπή Περίφ και στην, περι... και στην Επιτροπή Γιν φαίνεται ότι απορρίπτονται οι τροπολογίες μας συνέχεια. Αυτό με απογοητεύει γιατί προσπάθησα να εξηγήσω και στις δύο αυτές επιτροπές πόσο σοβαρά παίρνουμε το θέμα. Υπάρχει όντως ε, μια έλλειψη, σοβαρή έλλειψη στη συλλογή στοιχείων και στη δικτύωση των χωρών μελών θα έπρεπε εκεί να ζητήσουμε βελτίωση για υγειονομικούς δείκτες με βάση τα φύλλα. Υπάρχει δυνατότητα να ληφθούν νομοθετικά μέτρα, καμπάνιες ε, και ταύτιση των βελτίστων πρακτικών. Και νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε εμείς ιδιαίτερα ότι υπάρχει το θέμα των μειονοτικών γυναικών. Όσο για τα στοιχεία που ήδη υπάρχουν από επιστημονικούς οργανισμούς δείχνουν ότι οι γυναίκες στις μειονότητες είναι στη χειρότερη υγειονομική κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι θέλουμε η Επιτροπή Περίφ στη γνωμοδότησή της να το τονίζει και εκείνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Παρβάνοβα. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Φίγκερ εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαφώς ε, το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η υγεία είναι βασικό ζήτημα. Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Και φυσιολογικό είναι, επειδή οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά να έχουν και π.χ. έχουν τα ζητήματα της μητρότητας ε, δουλεύουν διαφορετικά συχνά έχουν δουλειές που επηρεάζουν την υγεία συχνά έχουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα Οπότε η υγεία είναι σημαντική για τις γυναίκες. Εν πάση περιπτώσει η υγεία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, η οικονομική και κοινωνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παίζει σημαντικό ρολό. Βλέπετε πως έρχονται πακέτα λιτότητας και αυτό επηρεάζει την υγεία των γυναικών και των πολιτών, αλλά ειδικά των γυναικών. Υπάρχουν προβλήματα με τις τιμές των φαρμάκων, με την πρόσβαση στις θεραπείες. Συχνά μόνο οι πλούσιοι έχουν πρόσβαση στην υγεία. αλλά νομίζω πως αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη γνωμοδότηση. <laughs> Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει εδώ πέρα πολύ χώρος. Συμφωνώ με αυτά τα οποία ακούστηκαν, αλλά πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να δούμε αυτά τα αισθήματα σε πιο μεγάλο βάθο. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σινκλέρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπαν και άλλοι, εδώ πρόκειται για δικαιοδοσία των χωρών μελών και πρέπει να παραμείνει τέτοια. Από ό,τι ξέρω εγώ για την υγεία, το φύλλο που είναι στη χειρότερη υγειονομική κατάσταση είναι οι άντρες. Αυτοί έχουν περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου και για αυτοί διστάζουν περισσότερο από τις γυναίκες να πάνε στο γιατρό. Αλλά παρόλα αυτά, πολλές από τις προτάσεις που έγιναν εδώ τις δέχομαι. Γενικά, όταν διαβάζει κανείς τέτοιες εκθέσεις, πρέπει να υπάρχει κάποια μεγαλύτερη αναγνώριση του γεγονότος ότι ζούμε σε συνθήκες λιτότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν γίνει μεγάλες περικοπές στο υγειονομικό, στον υγειονομικό τομέα. Πρέπει όμως να προσέχουμε γιατί συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυγχάνει όταν κάνει τα πράγματα πολύ γρήγορα και υπερβολικά ενώ η προσέγγιση βήμα προς βήμα είναι η πιο αποτελεσματική. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αν πιέσουμε υπερβολικά δεν καταλήγουμε πουθενά. Ορίστε τι γράφει ο Βασιλιακός τύπος. Ότι θα καταστεί παράνομο για τις ασφαλιστικές εταιρείες να αναλυθεί το φύλλο του ετούντος. Αυτό θα βλάψει τις γυναίκες διότι αυτή η υπερβολική πολιτική ισότητα των φύλων δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονό ότι δεν είναι ίσα τα φύλλα, δεν είμαστε το ίδιο γυναίκες και άντρε. και πρέπει να προσέχουμε πώς κάνουμε τις διατυπώσει μας εδώ μέσα. Ευχαριστούμε. Κυρία Τόμσεν, ναι θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε η τελευταία ομιλήτρια για την άνηση μεταχείριση κατά των ανδρών στον υγειονομικό τομέα. Είχα πάει σε μία διάσκεψη το καλοκαίρι και οι Γερμανοί, οι Γερμανίδες ερευνήτριες είχαν κάνει μια μελέτη που νομίζω τα αποτελέσματά της ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και έδειχνε ότι οι άντρες δεν έχουν και τόσο πολλά προνόμια, ότι 75% των οργάνων που δορίζονται προέρχονται από γυναίκες και οι περισσότεροι που εποφελούνται είναι άντρες. Τα πειράματα για τα φάρμακα γίνονται σε άντρες. Τα δίνουν μετά σε γυναίκες, πεθαίνουν πολλές και Γι' αυτό νομίζω ότι και για τις καρδιαγγειακές θεραπείες υπάρχει προνόμιο και προτεραιότητα δίνεται στους άντρες. Υπάρχουν πολλές ανισότητες εδώ. Ο κύριος Σοβέν, κυρία Πρόεδρε. Εδώ μιλάμε για ισότητα των φίλων και δικαιώματα των γυναικών. Με συγχωρείτε κυρίες μου, αλλά πρέπει να αναγνωρίσετε ότι η ανισότητα είναι υπέρ των γυναικών, μάλλον παρά υπέρ των ανδρών στον υγειονομικό τομέα. Γιατί το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι πολύ χαμηλότερο από των γυναικών. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό στοιχείο που δεν το αμφισβητεί κανείς και παρατηρείται σε όλες τις χώρες. Το θέμα που πρέπει να θέσουμε ίσως είναι με τα συγχωρήσεως να δούμε γιατί υπάρχει τέτοια ανισότητα. Δεύτερον, είπατε οι γυναίκες έχουν χειρότερη περίθαλψη. Ναι, αλλά αν οι γυναίκες έχουν λιγότερες εγχειρήσεις καρδιαγγειακές είναι γιατί έχουν λιγότερες καρδιαγγειακές παθήσεις. Γι' αυτό. Έτσι είναι τα πράγματα. Μα με συγχωρείτε κυρίες μου. Μπορεί να μην ξέρω πολλά πράγματα αλλά είμαι γιατρός και η ειδικότητα μου αυτή είναι η καρδιολογία. Ε, Τι να κάνω, αυτά σπούδασα. Λοιπόν, όλες οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η θνησιμότητα από καρδιαγκιακές παθήσεις αλλά και άλλες, Αλτσχάιμερ κλπ είναι μεγαλύτερη στους άντρες για διάφορους λόγους που δεν, θα τους, εξηγούν, τους εξηγούν πάντα, δεν τους ξέρουμε όλους, περιβάλλον, κάπνισμα κλπ. Αλλά πάντως είναι γεγονός. Οι άντρες έχουν περισσότερες εγχειρήσεις bypass γιατί έχουν περισσότερες παθήσεις. Αυτή η ανισότητα δεν είναι αγνοήσιμη. Αφού είμαστε και ισότητα των φύλων, επιτροπή και ισότητα των φύλων, πρέπει να μιλήσουμε και για τα δύο φύλλα. Τώρα, υπάρχουν ανισότητες και κατά των γυναικών και πρέπει να τις αναφέρουμε. Τις είπατε πολύ σωστά. Και σχετίζονται με κοινωνικούς παράγοντες. δεν είναι τόσο η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη που είναι κατά των γυναικών γιατί είτε είναι κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλούσιος είτε πτωχός υπάρχει περίθαλψη η δυσκολία έγκυται στις τρέχουσες θεραπείες δηλαδή όταν, στην πρόσβαση στον απλό παθολόγο όχι στις βαριές παθήσεις στα δόντια, στα μάτια εκεί υπάρχουν ανισότητες στην καθημερινή ζωή, παθήσεις της καθημερινής ζωής και τρίτον όταν κανείς έχει την ατυχία να ανήκει σε κοινωνικο-οικονομική κατηγορία μη προνομιούχα μπορεί να έχει περισσότερους να σημειώνονται περισσότεροι καρκίνοι ας πούμε να μην ψάχνουν τον καρκίνο της μήτρας όσο θα έπρεπε. Αλλά πρέπει να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Πρώτον, υπάρχει ανισότητα υπέρ των γυναικών και κατά των ανδρών στα υγειονομικά. Πρέπει να το πούμε και μέσα στις γυναίκες η διαφορά έγκυται στην κοινωνική διαφορά, στην κοινωνικο-επαγγελματική διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω εγώ πριν την κυρία Παρβάνοβα θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω το ότι πρέπει να θυμόμαστε πως οι γυναίκες ζουν πράγματι περισσότερο. Και πράγματι οι γυναίκες έχουν πολύ χειρότερη υγεία όσο ζουν. Οπότε πιο συχνά διαπιστώνουν οι γυναίκες ότι είναι άρρωστες. Πρέπει να ρωτηθούμε γιατί το αισθάνονται αυτό. Γιατί αισθάνονται ότι έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας. Δεν είναι μόνο το πότε πεθαίνει κανείς, αλλά και το τι συμβαίνει όσο ζει. Συμφωνώ με τον κύριο Ζωβά. Ξέρουμε πως η υγεία εξαρτάται από διάφορες μεταβλητές. Κοινωνικο-οικονομικές τα κτλ. Υπάρχει λοιπόν ανισότητα στην υγεία ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων. Αλλά μπορούμε να πούμε πως ε, υπάρχει ανισότητα και όσον αφορά το κόστος της υγείας. Το οποίο εξαρτάται από το φύλλο. Εγώ έχω δει κάποιες μελέτες που λένε σαφώς πως παραδείγματος χάρη που λένε. Παραδείγματο χάρη πως όταν τηλεφωνούμε στο ασθενοφόρο περιμένουν περισσότερο οι γυναίκες από του άντρε. Γιατί δίνουν προτεραιότητα στι γυναίκες. Στους άντρε με συγχωρείτε. Υπάρχουν τέτοιες μελέτες. Είναι σαφές, σαφές. σαφές. Το βασικότερο και το σαφέστερο είναι όταν έχουν την ίδια αρρώστια άντρας και γυναίκες. Εκεί πέρα φαίνεται πως 20% των του συνολικού κόστους της υγείας στη χώρα μου τη Σουηδία θα μειώνονταν το κόστος κατά 20% εάν μειώναμε το επίπεδο περίθαλψης, το επίπεδο που παρέχεται στις γυναίκες. Δεν θα σας απασχολήσω άλλο, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για την ίδια ασθένεια, π.χ. όταν έχουμε δερματολογικά προβλήματα ανδρών και γυναικών, οι γυναίκε του γράφουν μια συνταγή και του λένε πήγαινε στο φαρμακείο. Ενώ αν πάνε οι άντρες, τους δίνουν φωτοθεραπεία, που είναι πιο ακριβή. Οπότε βλέπετε η πιο ακριβή θεραπεία πάει στους άντρες. Αυτή δεν ήταν καμία μελέτη με άντρες γιατρούς όλοι οι γιατροί στη μελέτη ή εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι ήταν γυναίκες. Οπότε δεν είναι έτσι τόσο απλό το ζήτημα. Ας πάνω είναι ένα θέμα που θα ελπίζω να συνεχίσουμε να συζητάμε. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Παρβάνοβα παρακαλώ. Uh, <laughs> θα ήταν ένα μεγάλο λάθος εάν φτάσουμε σε μία ρήξη μεταξύ ε, των δύο φίλων, μιλώντας για το ποιος είναι σε πιο προνομιούχο θέση. Το θέμα αυτό πλήττει όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει διαφορετικό προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες και τις γυναίκες. Έχουμε 16 φορές περισσότερο φυματίωση σε ορισμένε χώρες, 6 φορές περισσότερους θανάτους από καρκίνο σε ορισμένα ε, κράτη-μέλη σε σχέση με άλλα. Ασχολούμαι για 20 χρόνια με θέματα υγείας και λαμβάνω το λόγο περισσότερο ε, ως εμπειρογνώμων. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερους δείκτες όταν, μεταξύ των δύο φίλων ως προς την ε, πιθανότητα να πληγεί κάποιος από μία ασθένεια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό έχει σχέση με τα εθνικά συστήματα υγείας και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών αφενός και επιπροσθέτως υπάρχει και το θέμα των δύο φύλων, υπάρχει και το θέμα ότι οι γυναίκες, ε, οι άνδρες είναι σε καλύτερη θέση, βεβαίως πλήττονται περισσότερο από καρδιοαγγειακά, αλλά οι γυναίκες, αυτό είναι ο πρώτος παράγον θανάτου για τις γυναίκες, δηλαδή. και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε συγκεκριμένα, να φτάσουμε σε συγκεκριμένους δείκτες για να μην μεροληπτούμε και ίσως φτάσουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα, δηλαδή θα φαίνεται ότι οι γυναίκες ή οι άνδρες έχουν καλύτερη πρόσβαση ή δεν την χάνουν της ίδιας ιατρικής προσοχής και ούτω καθεξής. Αυτό θα ήταν λανθασμένο. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών με βάση αποδείξεις και με βάση αυτούς τους μηχανισμούς θα δουν πώς θα δράσουν και πώς θα ε, ορίσουν μία εθνική πολιτική υγείας και μπορούν να φτάσουν στη μία ή στην άλλη προτεραιότητα και να φέρουν την ευθύνη ως κράτη-μέλη για την υγεία των πολιτών. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε στα εθνικά συστήματα υγείας, ούτε να έχουμε μία ρήξη μεταξύ των δύο φύλων. Απλώς να έχουμε μία καλύτερη ιδέα που υφίστανται τα προβλήματα και πώς μπορούν να πληρωθούν αυτά τα κενά. Περί αυτού πρόκειται. Ευχαριστούμε κυρία Παρβάνοβα. Ο κύριος Ζουβέ. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Συμφωνώ με την κυρία Παρβάνοβα, το θέμα είναι πολύ σημαντικό και επειδή προβαίνουμε σε μια κατάφαση δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και σωστή, θα πρέπει να αποδειχθεί. Συμφωνώ με την κυρία Σβένσα. Ας μου βρείτε αυτό το έγγραφο το οποίο δείχνει ότι οι γυναίκες έχουν μακροζωή μεγαλύτερη από τους άνδρες, αλλά έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής και υγείας και όταν έχουν, ε, ας πούμε, έχουν έξεμα, νομίζω ότι δεν υπάρχει η θεραπεία που είπατε, δηλαδή με τις ε, υπέρυθρες. Περιόδη. Η συγγνώμη. Και νομίζω δεν υπάρχει μια τέτοια θεραπεία. Το γεγονός ότι λέτε κάτι δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια. Eh, Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σεμάνσκι. Νομίζω ότι πολλές συζητήσεις, οι συζητήσεις μάλλον οδηγούν σε επιχειρήματα τα οποία δεν είναι και ε, απολύτως εύλογα ή σωστά. Υπάρχουν λίγοι άνδρες σε αυτή την Επιτροπή, υπάρχουν ε, πολλά αμφιλεγόμενα και όλα αυτά οδηγούν σε μία συζήτηση. Δηλαδή, είναι καλύτερα να έχουμε ε, μία καλύτερη ποιότητα ζωής παρά μακροζωία. Οι άνδρες δεν ζουν τόσο πολύ όσο οι γυναίκες αλλά αυτά τα επιχειρήματα δεν έχουν λόγο ύπαρξης πολλές φορές, δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερη η μακροζωία και ας μην είναι τόσο πολύ ποιοτική, ποιοτικά καλή. Αλλά αυτός, αυτός είναι ο βιολογικός κύκλος. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι οι άνδρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες γιατί μία μέση γυναίκα ε, ζει 73 ε, χρόνια, ενώ ε, ένας άνδρας 61. Και για να εξορροπήσουμε το συνταξιοδοτικό, προτάθηκε να αυξήσουμε το όριο συνταξιοδότησης στα 65 για τον Ρώσο άνδρα. Δηλαδή, ζει κατά μέσο όρο 61, ε, ας συνταξιοδοτηθεί στα 65. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να επικεντρωθούμε σε ζητήματα τα οποία δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Θα πρέπει να είμαστε πιο συμπονετικοί προς τους άντρες, να είσαστε δηλαδή. Και αυτό αφορά και την πρόεδρο. Θα πρέπει να το προωθήσει δηλαδή η η πρόεδρος και μπας το χιούμορ είναι το καλύτερο φάρμακο για όλα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιμάνσκι. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση σήμερα το πρωί. Έχει σημασία να έχουμε πολλές γνώμες, πληθώρα γνωμών και μιλάμε βεβαίως για ισότητα, ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και ε, γυναικών. Κυρία Σκοπά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη Ήμουν εκτός συζήτησης διότι έπρεπε να μεταβώ σε μία άλλη ε, επιτροπή. Αλλά από ό,τι καταλάβαλα συζητάτε για τα εθνικά συστήματα υγείας. Και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω σε σχέση με την πρόσβαση στον τομέα υγείας, στο σύστημα υγείας. Ε, ε, Ένα από τα άρθρα που προτείνουμε μιλάει για το προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, ότι θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Νομίζω όμως ότι οι γυναίκες βρίσκονται, κατέχουν μάλλον θέση νοσηλεύτριας, νοσηλεύτριας περισσότερα. Νοσηλεύτρια. Δηλαδή ε, δεν ανήκουν τόσο πολύ στο ιατρικό προσωπικό. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ίση εκπροσώπηση. Συγγνώμη, αλλά δεν βρίσκω το άρθρο, τον αριθμό. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Εστρέλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η συζήτηση είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Είναι, πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο που αφορά πολλούς τομείς. Είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας. Μιλάμε για αλληλεγγύη στον ε, τομέα υγείας, μείωση ανισοτήτων στον τομέα υγείας και αυτό σημαίνει αλληλεγγύη υπό όλες τις μορφές για όλα τα κοινωνικά στρώματα, για τα δύο φύλλα, για ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως ε, διάκριση. Στα πλαίσια της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης, οπωσδήποτε θα υπάρχει και επιδίνωση της πρόσβασης στα συστήματα υγείας. Υπάρχει δυσκολία πρόσβασης και αυτό αφορά και τα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα ελέγχθη ότι το προσδόκιμο ζωής, το μέσο προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και το μέσο προσδόκιμο είναι υψηλότερο για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες. Θα ήθελα όμως να πω ότι υπάρχει και ε, διαφορά μεταξύ προσδοκίμου μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ε, στρωματοποίησης. Δηλαδή υπάρχει διαφοροποίηση 10 χρόνων για τους άνδρες και 6 χρόνων για τις γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που ευημερούν ζουν και περισσότερα. Και οι άνδρες έχουν ε, πλεονέκτημα σε σχέση με τις γυναίκες. Βεβαίως ε, υπάρχουν οι μετανάστες, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, οι εθνοτικές μειονότητες, οι άστεγοι, αυτοί που αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα πρέπει να διορθώσουμε κάπως αυτές τις ανισότητες, να παρέμβουμε, να παρέμβουμε έτσι ώστε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι πολλαπλοί παράγοντες ως προς την εκπαίδευση, κατάρτιση, πρόσβαση στο σύστημα και ούτω καθεξής και γενικότερα διαφοροποιήσεις που υπάρχουν. Επίσης υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. και διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες έχουν χαμηλότερο μισθό από τους άνδρες, της τάξης του 18% και αυτό αποτελεί μειονέκτημα για τις γυναίκες ως προς την πρόσβαση στα εθνικά συστήματα υγείας. Ο κύριος Ζουβέν, ο οποίος αποχώρησε, αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα. Θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα και σε αυτούς που είναι γιατροί και σε εκείνους που δεν είναι. Τα καρδιοαγγειακά πλήττουν περισσότερο τους άνδρες και αυτό αφορά τον ε, βιολογικό κύκλο, ε, το DNA ή τον ε, τρόπο ζωής δηλαδή ότι οι άντρες ε, αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, ε, ζουν καλύτερα, έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, καπνίζουν, πίνουν, απολαμβάνουν τη ζωή τους. Πολύ περισσότερο από τις γυναίκες. Ε, άρα πεθαίνουν και νωρίτερα. Αλλά πεθαίνουν ευχαριστημένοι. Και αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να δούμε το προσδόκιμο ζωής αλλά να το εντάξουμε κάπου και κάπως καλύτερα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η κοινωνική και επαγγελματική πλαισίωση του ζητήματος. Εάν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, θα πρέπει η καταπολέμηση των ανισοτήτων αφορά όλους τους τομείς, έτσι ώστε να υπάρχει και καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας. Θα υποβάλω ορισμένε τροπολογίες στη γνωμοδότηση αυτή έκθεσή μου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας θα είναι έτοιμη για μετάφραση στις 8 Νοεμβρίου. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Και το 2011 θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια η έκθεση αυτή. Επειδή όμως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και χρειαζόμαστε και τη γνωμοδότηση της εσωτερικής αγοράς, αυτές οι συζητήσεις στις ε, διάφορες επιτροπές θα εμπλουτίσουν το περιεχόμενο και ιδιαίτερα για μένα ως εισηγήτρια επί της Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Εστρέλα. Θα περάσουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω λόγο στον κύριο Φανόρχαιμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά. Ε, υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες εδώ, πολύπλοκες και δυσκολίες. αλλά πάντα μπορεί κανείς να υποφεληθεί μαθαίνοντας. Η Κομισιόν διδάσκει αίγε, διγεράσκει αίγε διδασκόμενη. Λοιπόν, πάντοτε πρέπει να βάζουμε την κοινωνική διάσταση. Δεν είναι μόνο η διαφορά των φίλων αλλά και οι κοινωνικές διαφορές. Θα ήθελα να πω ότι Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ανακοίνωσης είναι ότι προσπαθεί να μας μάθει ποιες πολύπλοκες σχέσεις υπάρχουν μεταξύ βιολογίας και περιβάλλοντος. Και νομίζω καλό θα ήταν για όλους να, γνωρίζει ότι, να, γνωρίζουν ότι η διαφορά του προσδοκίμου ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι η ίδια παντού. Και αλλάζει στις χώρες που έχουμε τα περισσότερα στοιχεία τουλάχιστον και πρόκειται για θέμα κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων. Από τις μετρήσεις που έχουμε για τα φύλλα βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή ισότητα ως προς τις ασθένειες και την επιβίωση. Οι διαφορές των φύλων δεν είναι απλώς βιολογικές σε αυτό το θέμα. Και εδώ το όλο θέμα είναι να μάθουμε όλοι να καταλάβουμε τη σημασία που έχουν κοινωνικές πτυχές και οι σοβαρότεροι από αυτές είναι ίσως οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και το περιβάλλον. Επίσης, όλες αυτές οι μεταβλητές ξεπερνούν κατά πολύ το απλό τους άθροισμα γιατί το εκπληκτικό είναι ότι σε ολόκληρη την κοινωνική ιεραρχία παρατηρούνται ανάλογα φαινόμενα. Ένας ανώτατος υπάλληλος της Κομισιόν μπορεί να έχει χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής από έναν πιο χαμηλό βαθμό υπάλληλο. Αυτό δείχνει ότι γενικά κατά μέσο όρο συνολικά οι ευκαιρίες που έχουμε στην κοινωνική ζωή αντικατοπτρίζονται τελικά και στο προσδόκιμο ζωής μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Ταραμπέλας. Κύριε Πρόεδρε, όλα υπόθηκαν. Φαίνεται ότι τελικά το στρες είναι ο καθοριστικός παράγοντας και ίσως οι άντρες ζουν λιγότερο γιατί ζουν μεγάλη αγωνία κατά τους αγώνες ποδοσφαίρου. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω σε αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι υπάρχει εδώ και ο δετερμινισμός των κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων. Ο κύριος Σοβέν μας είχε πει ότι στις βαριές παθήσεις που απαιτούν νοσηλεία μπορεί να υπάρχουν διαφορές αλλά όλοι την χάνουν περίθαλψης. Αντίθετα στις καθημερινές παθήσεις και άρα στις λιγότερο σοβαρές νοσηλίες οι άντρες πηγαίνουν λιγότερο στο γιατρό ε, χρησιμοποίησε το παράδειγμα των οδόντων αλλά το ίδιο συμβαίνει και για τη διατροφή δεν προσέχουν τη διατροφή τους τρώνε πράγματα που θεωρούνται πιο εύκολα αν και δημιουργούν παχυσαρκία ιδιαίτερα στους νέους αυτό το φαινόμενο αυξάνεται και άρα εδώ στη διατροφή πρέπει να τονίσουμε περισσότερο το θέμα μεγαλύτερης δικαιοσύνης στην πρόληψη από την οικογένεια ήδη και από το σχολείο βέβαια. Πολύ ωραία, ήταν ζωηρή και ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Η διορία κατάθεση τροπολογιών λίγη στις 10 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 29 και 30 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή περίφου που είναι αρμόδια επί της ουσίας τέλη Ιανουαρίου. Τώρα επόμενο σημείο. Επόμενο σημείο. Η, πράσινη, η γνωμοδότηση για, την πράσινη, για μία πράσινη βίβλο της Κομισιόν για ένα επαρκές και βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα. Για μας αρμόδια είναι η κυρία Ματέρα. Ε, ήθελα λοιπόν τώρα να ζητήσω την κυρία Ματέρα να μας κάνει μια εισαγωγή. Έχετε το... Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πράσινη βίβλο για τα συνταξιοδοτικά στην Ευρώπη. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό με βάση τη γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού και την μείωση των γεννήσεων. Ε, είναι πολύ φιλόδοξο αυτό το σχέδιο και στην Πράσινη Βίβλο υπάρχουν πολλές υποδείξεις, κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών, τη μεταρρύθμισή τους, διότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά αρμοδιότητες καθαρά κρατικές. Υπάρχουν όμως και βασικοί μηχανισμοί για να περιορίσουμε κατά το δυνατόν τα εμπόδια που καθιστούν αδύνατη την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, έτσι ώστε να μας ενδιαφέρει καθε η κινητικότητα των εργαζομένων, γιατί πολλές φορές οι εργαζόμενοι απαρνούνται μία σταδιοδρομία όταν θα πρέπει να διασχίσουν τα σύνορα, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς ε, των δικαιωμάτων από το ένα κράτος στο άλλο. Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Γυναικών θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε την ανισότητα σύνταξης, συνταξιοδοτικού, ως προς τους άνδρες και τις γυναίκες. Ξέρουμε ότι υπάρχει ε, ένα μισθολογικό χάσμα της τάξης του 17% μεταξύ ανδρών και γυναικών, άρα οι γυναίκες έχουν και χαμηλότερες συντάξεις. Επίσης, οι γυναίκες γυναίκες επιλέγουν επισφαλή εργασία ή μερική εργασία για να ασχοληθούν με παιδιά, με ασθενείς ή με γυρεότερα μέλη της οικογένειας και αυτό σημαίνει ότι έχουν και χαμηλότερες συντάξεις. Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες εκτίθενται σε περισσότερους παράγοντες φτώχειας γιατί έχουν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε και θα πρέπει να κάνουμε μία προβολή για ίση συνταξιοδότηση, ίσα δικαιώματα με βάση μία αναλογιστική μελέτη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά, με του, τα πλέον ασθενή μέλη της ε, οικογένειας και τα γυρεότερα. Επίσης, γι' αυτό πιστεύω ότι θα έχουμε μία εξαιρετική έκθεση και από πλευράς ε, Επιτροπής Απασχόλησης. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Τσέσκοβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Τώρα θα συζητήσουμε μια έκθεση η οποία εγώ νόμιζα βέβαια ότι θα συζητούν νωρίτερα. Έχω μια παρατήρηση στο σημείο Δέλτα που λέει ότι οι γυναίκες και οι άντρες πρέπει να είναι ίσοι όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης στην Τσεχία οι γυναίκες έχουν πλεονέκτημα. Γιατί βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη και λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των παιδιών όταν υπολογίζουν την ηλικία συνταξιοδότησης. Ε, και βεβαίω οι γυναίκες, ε, ε, αν ισχύσει αυτό, θα χάσουν το πλεονέκτημα αυτό που έχουν στην Τσεχία. Επιπλέον, έχω ένα ερώτημα για το σημείο 3, που λέει ότι ε, υπόψη ε, πω ιδιότερα τα νέα κράτη-μέλη πρέπει να αναθεωρήσουν ε, τα συνταξιδοτικά συστήματα λαμβάνοντα υπόψη το ότι οι γυναίκε ζουν περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, πώ να το ερμηνεύσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τον κύριο Σιμάνσκι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα εγώ να επισημάνω ένα ζήτημα που αφορά τον κοινωνικό και οικογενειακό ρόλο των γυναικών όσον αφορά παραδείγματος χάρη την ανατροφή των παιδιών. Στην Τσεχία πράγματι αυτό το οποίο κάνουμε νομίζω πως μπορεί να αποτελέσει έμπνευση. Ε, και θεωρώ πως η Επιτροπή μας πρέπει να αποφύγει τη διακριτική μεταχείριση των γυναικών γιατί αναλαμβάνω ειδικά αν σκεφτούμε τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ξαναλαμβάνονται λαμβάνονται πολλές δράσεις ε, με στόχο να αποφευχθούν τα δημογραφικά προβλήματα. Οπότε θεωρώ πως αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν σοβαρά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως σε πολλά κράτη-μέλη τα ζητήματα, τα συστήματα υπολογισμού των συντάξεων είναι διαφορετικά. Συχνά οι γυναίκες ε, κερδίζουν λιγότερα, δουλεύουν λιγότερες ώρες και ζουν περισσότερο. Γι' αυτό έχουν μικρότερη συντάξη. Ενώ οι άντρες δουλεύουν περισσότερο, βγάζουν περισσότερα και ζουν και λιγότερο. Οπότε παίρνουν σύνταξη για λιγότερο χρόνο. Και συχνά χρησιμοποιούμε αυτό το σταθμισμένο μέσο όρο για τον υπολογισμό των συντάξεων και αυτό οδηγεί στο να είναι υψηλότερε οι συντάξει των γυναικών από τις εισφορέ που έχουν πληρώσει. <clears throat> και σε πολλές τέτοιε περιπτώσεις πρέπει να παρέμβει το κράτος. Δηλαδή, αυτό είναι θέμα του πώς αντιλαμβανόμαστε την ισότητα στην αγορά εργασίας. Δεν φταίνει οι άντρες που δουλεύουν περισσότερο και ζουν λιγότερο. Μιλάμε για διακριτική μεταχείριση εις βάρος των γυναικών. Οπότε είναι πολύ θετικέ αυτές οι διατάξεις. Ελπίζω να μείνουν και να συμπληρωθούν με βάση το τσέχικο παράδειγμα. Εξάλλου γυναίκες εργάζονται σκληρά στο σπίτι ε, και φροντίζουν την οικογένεια. Η γυναίκα συνεισφέρει στο ΑΕΠ και δεν λαμβάνεται υπόψη. Και συχνά τιμωρείται τον τελειώσει ε, επαγγελματικό της βίο Πρέπει να στηριχθεί από το κράτος ή από κάποιον που έχει σύνταξη. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Μπόιτοβα. κυρια μποιτοβα ευχαριστω να αναφέρθω σε αυτό το οποίο είπε ο Τσέχος συνάδελφος. Βεβαίω, κάθε χώρα χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σύστημα για να υπολογίσει και να λάβει υπόψη την φροντίδα των παιδιών όταν ε, υπολογίζεται η ηλικία της συνταξη. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε το να μειώσουμε αυτό το οποίο είχαν επιτύχει ορισμένες χώρες με το να εξισώσουμε τα όρια. Θεωρούμε πως η μητρότητα και η φροντίδα των παιδιών πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάθε χώρα πρέπει να βρει έναν τρόπο να το οργανώσει. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να εξετάσουμε είναι γεγονός πως φαίνεται περίεργο όταν οι γυναίκες ζουν περισσότερο να βγαίνουν και νωρίτερα στη σύνταξη. Αλλά υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, εάν η γυναίκα φροντίζει τα παιδιά για πολλά χρόνια, αν έχει πολλά παιδιά παραδείγματος χάρη, μπορεί να συμβεί το εξής. Ο αριθμός ετών που ε, δούλεψε να είναι χαμηλότερος και άρα θα τις ε, ζητούσα να συνταξιοδοτηθεί αργότερα από τους άντρες. Γι' αυτό πρέπει να σχετίζεται με τον αριθμό των παιδιών. Και βεβαίως ότι οι άντρες ε, πεθαίνουν νωρίτερα είναι δικό τους πρόβλημα. Εάν φρόντιζαν περισσότερο τα παιδιά και ήταν πιο υγιείς, ήταν καλύτερα. Κύριος, κύριε Παπαδοπούλου. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και διακοιμάσεις όσον αφορά τα συνταξιδοτικά συστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Και οπωσδήποτε ο αναλογιστικός υπολογισμός των συνταξιδοτικών συστημάτων βασίζεται κυρίως στο μισθό και στις εισφορές κατά την περίοδο εργασία. Είναι κάπως ε, παλιά συστήματα τα οποία υιοθετούνται και πολλές φορές χρειάζεται εξυγχρονισμός ιδίω στι μέρε μα που η γυναίκα έχει μπει δυναμικά σε αρκετέ χώρε στην αγορά εργασία, ενώ αλλού χρειάζεται κίνητρα για να μπει στην αγορά εργασία. Οπωσδήποτε αυτή η αναθεώρηση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την ανάγκη για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανισότητες όσον αφορά τις αμοιβέ ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες το γεγονός ότι οι γυναίκες συνήθως απασχολούνται σε επισφαλής ή μερικής απασχόλησης θέσεις εργασίας. Το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι πιο εκτεθειμένες λόγω στερεοτύπων και λόγω διακρίσεων σε δυσμενεί συνθήκε εργασίας και πολλές φορές ε, ζουν κατά από το όριο της φτώχειας, ειδικά οι γυναίκες μονογονεί ή γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη το μισθολογικό χάσμα. Έχει αναφερθεί προηγουμένως από την κυρία Ματέρα και από άλλους ότι αυτό το χάσμα κυμαίνεται από 17% μέχρι και 20%, πολλές φορές φτάνει και στο 23%. Ε, επίσης, το προσδόκιμο όριο των γυναικών ε, το προσδόκιμο όριο ζωή είναι ψηλότερο από αυτόν των ανδρών. Πολλέ ηλικιωμένε γυναίκε, οι οποίε ζουν μέχρι τα 78, τα 80, τα 85 χρόνια, αναγκάζονται ακριβώ να παίρνουν μια σύνταξη που είναι πολύ χαμηλή και δύσκολα μπορούν να ξεπεράσουν προβλήματα τη καθημερινότητα. Επομένω, εμεί προσβλέπουμε στο να γίνει ακριβώ μια αναθεώρηση, να υπάρχουν μίνιμουμ συνταξιοδοτικέ ε, ποσά για συντάξει, που να υποφελούνται όλες οι γυναίκες και οπωσδήποτε προσβλέπουμε ότι θα μπουν κατάλληλα και βιώσιμα κριτήρια, λαμβάνοντα σοβαρά υπόψη το κριτήριο του φύλου. Έχουμε αρκετέ ε, τροπολογίε τι οποίε θα προτείνουμε, ώστε να προσαρμοστεί και στην ιδεολογία τη Προδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, πάντα με στόχο ε, να συνυπολογιστούν όλε αυτέ οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε και η πράσινη βίβλος πιστεύω ότι παρέχει μια πολύ γερή βάση για να έχουμε επαρκή βιώσιμα και ασφαλή συνταξιδοτικά συστήματα, τα οποία με δικέ μα τροπολογίε θα γίνουν ακόμη καλύτερα για τι γυναίκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα εδώ πέρα να σας υπενθυμίσω πω έχουμε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Να ξεκινήσουμε. Γιατί έχουμε και 11.30 ώρα συνεδρία συντονιστών. Λοιπόν, ώστε να σχολιάσουν παρακαλώ να είναι σύντομοι. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ. Ε, είναι ένα ζήτημα συναρπαστικό να αναφέρω πως ε, οι ίσες ευκαιρίες καμιά φορά ε, έχουν και μειονεκτήματα. Με βάση αυτή την αρχή, το προνόμιο που υπάρχει ακόμα στο τσεχικό σύστημα όσον αφορά τις συντάξεις τερματίστηκε στη Σλοβακία γιατί τους έδιναν ε, μισό της εκατό για κάθε παιδί που ε, είχαν. Αλλά από την άλλη θυμάμαι πάρα πολύ καλά πως ε, υπήρχε μια απόπειρα να γίνει μια διαφορετική ένας διαφορετικός υπολογισμός των συντάξεων σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής ε, και την ηλικία συνταξιοδότησης. Δηλαδή υπήρχε μια διαφορά 7 ετών τότε. Οπότε το να δεχτούμε αυτές τις διαφορές στο νομικό σύστημα είναι πολύ επικίνδυνο Οπότε είναι δύσκολο για την Μπάρμπαρα να δημιουργήσει ένα τέτοιο συμβιβασμό. Η τροπολογία που θα αντανακλά όλες αυτές τις ε, διαφορές. Ε, αντιλαμβάνω πως ένα, έχουμε ένα ψήφισμα που υιοθετήθηκε το 2006, 2008, που αφορούσε το χάσμα αυτό στις πληρωμές των δύο φύλων γιατί είναι σαφές πως η διαφορά στις συντάξεις ανδρών και γυναικών σε μεγάλο βαθμό οφείλεται από τη διαφορά στις πληρωμές. Οπότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ η κυρία Λούλινγκ παρακαλώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη γιατί ήμουν απασχολημένη με άλλα ε, ζητήματα. Είμαι κοσμήτορ και είχα να ανταποκριθώ σε άλλα καθήκοντα. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Ματέρα. Όταν προβάλλουμε διεκδικήσεις θα είμαστε πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές ως προς τα, τα συστήματα στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω γιατί μιλάμε για αναλογιστικές μελέτες εδώ. Είναι μεν σημαντικές, αλλά δεν θέλετε να πείτε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτούς τους υπολογισμούς για να υπολογίσουμε τη σύνταξη. Διότι στη δική μου χώρα, όσο περισσότερο έχετε εργαστεί, τόσο περισσότερο υψηλότερος είναι ο μισθός και έχετε και υψηλότερη σύνταξη, διότι τι πληρώνουμε εισφορές με βάση το μισθό. Εκείνοι λοιπόν που εισέφεραν περισσότερο έχουν υψηλότερη σύνταξη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν όταν λέμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη μερική απασχόληση σε ένα σύστημα όπου η σύνταξη χρηματοδοτείται από τις εισφορές με βάση το δηλωμένο μισθό, δεν μπορείτε να ζητήσετε κάποιος που δούλεψε 8 ή 20 ώρες την εβδομάδα να έχει την ίδια σύνταξη με κάποιον που, διάβασε, που συγγνώμη, εργάστηκε 40 ώρες και εισέφερε και πλήρωσε τις εισφορές του. Μπορούμε να μιλήσουμε για ελάχιστες αποδόσεις, για ελάχιστη σύνταξη, για εκείνους που δούλεψαν λίγες ώρες. Εμείς έχουμε έναν ελάχιστο μισθό, αλλά είναι κάπως άδικο αυτό που θα πρέπει να υποστηρίξουμε είναι την εκπαίδευση. Ξέρω ότι τώρα το αποκτήσαμε, αλλά με τις εξοικονομήσεις που γίνονται θα το ξαναδούμε. Αυτό, αυτό είναι το πιο σοβαρό για τις γυναίκες, διότι χρειάζονται χρόνια εκπαίδευσης έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα ελάχιστο χρόνο δικαιοδότησης, δηλαδή απόκτησης δικαιώματος προς σύνταξη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν διατυπώνουμε τις ε, διεκδικήσεις μας. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Αυτή η πράσινη βίβλος ε, συνεγράφει, διότι προσπαθούμε να δούμε σημεία που διασυνδέονται μεταξύ τους. Εμείς θέλουμε μία ολιστική προσέγγιση για τη συνταξιοδότηση. Η Επιτροπή δεν έχει καμία πρόθεση να προβεί σε κατακαιρματισμό ή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε αυτό που κάνουμε έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται αυτές οι αλλαγές και στο, και στο συνταξιοδοτικό τη στιγμή που η υπογεννητικότητα είναι ένα στην ουσία υπάρχον σενάριο. Το Διευθυντήριο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα ασχοληθεί με το θέμα της ισότητας των φύλων ως προς το συνταξιοδοτικό και όταν έχουμε και τη δική σας έκθεση το Διευθυντήριο θα ορίσει την άποψή του υπομορφή λευκής βίβλου. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ματέρα. Έχουμε ακόμα δύο θέματα που θα μας απασχολήσουν. Και εγώ κοίταξα την ώρα και νομίζω ότι θα πρέπει να σας πω μία πρόταση. Έχει δει ο κυρία Λούλινγκ, ε, λέει ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Σύστημα το οποίο κατακαιρματίζεται σε 27 υπάρχουν πιο ασφαλή συνταξιοδοτικά συστήματα, γι' αυτό η Επιτροπή θα μπορούσε να βασιστεί εκεί για να προωθήσει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων θα ήθελα να έχω λίγη περισσότερη ώρα στο μέλλον, διότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να απαντήσω σε όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε πολύ. Στις 10 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε, έχουμε, μάλλον είναι η προθεσμία και 29 και 30 θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η γνωμοδότηση για τον ε, κανονισμό του Συμβουλίου σε σχέση με το διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό. Η κυρία Κλάς έχει το λόγο. Και έχουμε και μία επόμενη έκθεση. Η κυρία Νίμπλερ είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Αντικαθιστώ την κυρία Νίμπλερ η οποία σήμερα είναι σε συνέδριο του κόμματος στη Βαβαρία, στο Τσέσου γιατί είναι μέλος της ποσόστοσης των γυναικών στο Προεδρείο. Η έκθεση για τη θέση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και στην ε, διάσταση θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Σήμερα μιλάμε για 300.000 γάμους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είναι μεικτοί, δηλαδή προέρχονται οι έγγαμοι από διαφορετικά κράτη. Δυστυχώς όμως 140 με 170.000 αυτών των γάμων διαλύονται και λόγω βεβαίως των διαφορετικών διατάξεων περί διαζυγίου στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και με στόχο να διαμορφώσουμε ένα χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και δικαίου σε σχέση με την ε, ελευθερία των ατόμων θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όταν συγκρούονται οι διατάξεις για να δούμε ποιο το, θα είναι το δίκαιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Η κυρία Νίβλερ έχει συντάξει μια σύντομη έκθεση και θα ήθελα να τοποθεθεί σε διάφορες τροπολογίες. Η ένα είναι μια συμπλήρωση στο εκτιμώντας 16, όπου λέει κατά την πιστοποίηση επιλογή του δικαίου, οι σύζυγοι πρέπει να ενημερώνονται για τις νομικές συνέπειες που έχει η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου για να διασφαλίσουμε πως αυτό είναι σαφές και πως γνωρίζουν επακριβώς αυτές τις συνέπειες προβλέπει μία συμβολεογραφική πράξη της επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου η οποία θα αναφέρει και τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Επίσης θα πρέπει να μπορεί να υπάρχει μία βοήθεια για τα δικαστικά έξοδα. Ξέρετε πως υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις για τα δικαστικά έξοδα για να ληφθεί αυτό υπόψη αλλά και να διασφαλίσουμε πως ε, όπου υπάρχουν αυτές οι διατάξεις θα εφαρμόζονται κιόλας θέλουμε η χρήση αυτών των διατάξεων και σε διαζύγιο και σε περίπτωση διάστασης να ισχύει αυτό για να διασφαλιστεί πως ειδικά οι σύζυγοι εκείνοι οι οποίοι είναι ασθενέστεροι οικονομικά θα λαμβάνουν βοήθεια για τα δικαστικά έξοδα για να μην βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της οικονομικής τους ε, θέσης. Έχει να υπάρχει κοινός λογαριασμός στον οποίο τα υλικά να μην έχουν πρόσβαση, τέτοια πράγματα. Παραγραφή 2 και 5, αιτιολογική σκέψη 17, μιλάμε για μια γραπτή συμφωνία για την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης. Εκεί πέρα δεν επαρκεί αυτό, μια απλή συμφωνία. Μιλάει, όπως σας είπα, για πιστοποίηση με συμβολεογραφική πράξη. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια ηλεκτρονική μετάδοση συμβολιογραφικής ε, πράξης ε, για να μην ε, υπάρχει δυνατότητα παραποίησής της. Επίσης, για να λαμβάνω υπόψη τα διαφορετικά νομικά συστήματα, όσο δεν υπάρχουν κοινέ ρυθμίσεις, θεωρεί η εισηγήτρια πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς κανόνες ε, του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής τους. Και τέλος στο σημείο 4 μιλάμε για την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Στην πρόταση της Κομισιόν το πεδίο εφαρμογής μιλάμε μόνο για διαζύγιο και διάσταση. Η δε λύση γάμου δεν αναφέρεται, αντιθέτως αποκλείεται ρητά. Και σε κάποιες χώρες αυτό σημαίνει πως δεν ε, θεωρείται ότι είναι διαζευμένος κάποιος εάν δεν έχει λυθεί επισήμως ο γάμος. Οπότε θα πρέπει να, να ισχύει και στην περίπτωση στην οποία υπάρχει λύση του γάμου. Αυτά για αυτά τα οποία έχει προτείνει η κυρία Νίμπλερ και ευχαρίστω να ακούσω και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστούμε κυρία Κλάση, κυρία Παπαδοπούλου. Και σας παρακαλώ σύντομα. Actually, Mrs. President, I have uh, some questions from Mr. Έχω ορισμένε ερωτήσεις για τον κύριο Ταραμπέλα ο οποίος δεν είναι εδώ. Μία ερώτηση είναι προς την κυρία Νίμπλερ. Πρόκειται για τη δήλωση που μόλις ε, κάνατε. Δηλαδή, την επέκταση μέχρι την ε, ακυρότητα του γάμου. Ο κύριος Ταραπέλα ρωτά γιατί έχει, εφόσον έχει συμπεριληφθεί, στη συνέχεια ζητείτε από την τροπολογία να μην ληφθεί υπόψη. Μιλάμε για τη λύση του γάμου. Σε σχέση με το άρθρο 5, θα μπορούσατε να μας πείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Να ορίσετε την αρχή του lex fori Αλλά στην περίπτωση της Μάλτας που δεν αναγνωρίζει το διαζύγιο, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα ορισμένες επεξηγήσεις. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιες νομοθεσίες δεν προβλέπεται το διαξίδιο. Δηλαδή, όταν ε, δεν προβλέπεται η λύση του γάμου και το διαζύγιο. Επίσης, θα μπορούσατε να μας πείτε τι είναι ασύμβατο σε σχέση τι είναι ασύμβατο με το νόμο όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 επί του θέματος. Ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Πολύ σημαντικό το θέμα κυρία Πρόεδρε. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να παρέμβουμε πρέπει να δώσουμε κάποιο χρόνο γιατί είναι λεπτό το θέμα. Εγώ δέχομαι αυτή την πρωτοβουλία της Κομισιόν διότι εδώ και 45 χρόνια έχω ρωτήσει, έχω ζητήσει από την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα και ο τότε κύριος Αλτστάιν μου είχε πει ότι δεν είχε τη δικαιοδοσία διότι δεν το επέτρεπε τότε η συνθήκη. Και είχαμε τεράστιο πρόβλημα, ιδιαίτερα ως προς τον τουρισμό των διαζυγίων στην Ευρώπη, λόγω της διαφοράς των νομοθεσιών. Θέλω όμως να υπενθυμίσω ότι με δική μου πρωτοβουλία το 1995 είχαμε κάνει έκθεση πρωτοβουλίας για το splitting των δικαιωμάτων ε, διατροφής σε περίπτωση διαζυγίου και, ή συντάξεως. Και είχαμε πει θα καταθέσω ορισμένες τροπολογίες σύμφωνα με αυτά που είχαμε πει. Είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, να δούμε τι έχουμε ήδη ζητήσει από την Κομισιόν εδώ και 15 χρόνια δεν αντέδρασε, δεν έκανε τίποτε από όσα ζητήσαμε για να αποφευχθεί ο διαζευκτικός τουρισμός. Διότι στη Γερμανία υπάρχει το splitting των δικαιωμάτων σε περίπτωση διαζυγίου, ενώ σε άλλες χώρες όχι. Για να αποφευχθεί λοιπόν η μοιρασιά με γυναίκες που, των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων με γυναίκες που δεν έχουν ποτέ εργαστεί πηγαίνουν και ζητάνε διαζύγια στην από τη Γερμανία. Συμφωνώ ότι το θέμα είναι άκρο σημαντικό, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε μία προσκεκλημένη για το επόμενο θέμα. Κυρία Έσκοβα, να είσαστε ιδιαίτερα σύντομοι. Σύντομα. Θεωρώ πως είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα και χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο να το συζητήσουμε. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να εξηγήσουμε. Το πώς δηλαδή το ιδιωτικό δίκαιο των κρατών μελών θα χρησιμοποιηθεί Υπάρχουν πολλές νομικές στοιχείες που πρέπει να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αλέξης και από την Κομισιόν. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που προσκαλέσατε την Κομισιόν στη συνεδρίαση αυτή. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, την εισηγήτρια για το ότι τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά συνέταξε αυτή τη γνωμοδότηση. Συμφωνούμε με τη φιλοδοξία της Προεδρίας να τελειώσει ως το πιο σύντομα το θέμα αυτό και νομίζω πως ε, συνεισφέρει η Επιτροπή και εκτιμούμε πράγματι τις προσπάθειές σας. Έτσι διατηρείται ένας ρυθμός μετά την ε, απόφαση την που μας εξοδότησε τον Ιούλιο. Και όλοι θέλουμε να τελειώνουμε εδώ πέρα. Δεν θα μακρηγορήσω, θα περάσω στα ερωτήματα της κυρίας Παπαδοπούλου. Πρώτα απ' όλα, το πεδίο εφαρμογής του μέσου αυτού, γιατί εξαιρέθηκε η λύση του γάμου. Γιατί η λύση του γάμου σχετίζεται με ζητήματα ισχύως και ύπαρξης του γάμου. Εδώ μιλάμε για διαζύγιο όμως και διάσταση. Η λύση του γάμου θα πρέπει να μείνει εκτός. Αλλά δεν λειτουργούμε σε νομικό κενό. Υπάρχει ήδη ο κανονισμός Βρυξελών 2 που αφορά την πλήση του γάμου. Το ζήτημα είναι εδώ πέρα το εφαρμοστέο δίκαιο, δηλαδή με ποιο δίκαιο θα εκδικαστεί η υπόθεση όταν φτάσει ενώπιον ε, αρμοδίου δικαστηρίου σε κράτος μέλος. Σημείο 2. Η φύση του άρθρου 5. Το άρθρο 5 έχει συνταχθεί ως κανόνας εφαρμοστέου δικαίου που θα πρέπει να διακριθεί από τις γενικές ε, ρήτρες ε, πολιτικής στο άρθρο 7. Ε, έχει συμπεριληφθεί κατόπιν ετήσεως κάποιων κρατών μελών που είχαν εμπειρίες με αυτούς τους κανόνες εφαρμοστέου δικαίου για να αποφύγουμε, όπως μας είπαν τα κράτη-μέλη, το να περάσουμε σε χρονοβόρες διαδικασίες στα δικαστήρια. Κάποια δικαστήρια δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις ε, δημόσιας τάξης, οπότε κάνουν μία σύντομη εξέταση, λένε πως ε, λειτουργεί πάρα πολύ καλά στο σύστημα αυτό και συμφωνούμε με αυτό ως Κομισιόν. Η πρότασή μας του Μαρτίου προσπάθησε να ακολουθήσει την εντολή που μας έδωσαν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουμε με αυτή την πρόταση και αναλόγως να συμπεριληφθεί η πρόταση αυτή που υπήρχε ήδη στην συμβαστική πρόταση του 2008. Τρίτη ερώτηση. Τι σημαίνει σαφώς ασύμβατο με την δημόσια τάξη. Αυτή είναι μια ρήτρα που υπάρχει σε όλα τα μέσα εφαρμοστέου δικαίου δεν χρησιμοποιείται μόνο σε αυτό το, το δίκαιο της Ένωσης υπάρχει και στην Χάγη αλλά βεβαίως η δημόσια τάξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση στην Ένωση που έχουμε κοινή τον κοινό χώρο δικαιοσύνης πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των συστημάτων αυτών οπότε όταν λέμε εμφανώς, δηλαδή κανονικά εννοούμε πως πρέπει να τηρείται ο νόμος χωρίς προβλήματα και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να καταφεύγει σε αυτό το δικαστήριο. Κάποια άλλα σχόλια για την βιασύνη. Να σας πω πως η υπόθεση αυτή ξεκινήσε από το 2006 Έχουμε και κάποιες διατάξεις εδώ πέρα από την αρχή πρώτα του 2006 μετά από πρωτοβουλία των κρατών μελών. Η ενισχυμένη συνεργασία δεν είναι κάτι που μπορεί να προτείνει ε, η Κομισιόν. Είχαμε λίγο χρόνο να το σκεφτούμε. Πάντα πιέζει το χρόνο-διάγραμμα αλλά όπως σας είπα, ε, νομίζω πως η Επιτροπή σας ε, τα πάει καλά, συνεισφέρει και θα ήθελα να σας ζητήσω να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε ως το δυνατόν πιο σύντομα. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τα σχόλια αυτά. Ακούσουμε τώρα τα τελευταία σχόλια της κυρίας Κλάς. Ναι, σύντομα. Ευχαριστώ για τα σχόλια και για την αντιμετώπιση. Βεβαίως θα τα διαβιβάσω αυτά στην κυρία Νίμπλερ και πράγματι λείπει το τι γίνεται στις χώρες στις οποίες δεν υπάρχει διασυγείο, και στη Μάλτα δηλαδή αλλά πρέπει να δούμε ποιες, ποιες δυνατότητες έχουμε να τις γνωρίζουμε. Το θέμα εδώ είναι η ενισχυμένη συνεργασία και είναι πολύ σημαντικό αυτό να υπάρχει δηλαδή πληροφόρηση και να μην... Ε, δεν σημαίνει αυτό πως υπάρχει διακριτική μεταχείριση, αλλά πρέπει να ενημερώνεται κανείς ποια δικαιώματα έχει κάποιος και με ποιο δίκαιο παντρεύεται και με ποιο δίκαιο μπορεί μετά να ε, διαλυθεί ο γάμος. Νομίζω πως αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος. και τώρα για τα μονομένα ερωτήματα θα τα δει η κυρία Νίμπλερ και νομίζω θα οδηγηθούμε σε μια καλή συμφωνία στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κυρία Κλάση. Λοιπόν, πρέπει να βιαστούμε τώρα. Το επόμενο σημείο σε ημερήσια διάταξη είναι... Ε, α, να σας πω πως η προθεσμία τροπολογίας είναι 8 Νοεμβρίου, θα συζητηθεί στην Επιτροπή 29 και 30 Νοεμβρίου και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα το ψηφίσει 2 Δεκεμβρίου. Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο. Αφορά τον ρόλο των γυναικών στη Γεωργία και τις αγροτικές περιοχές. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Γέγκλε, Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο κυρία Γέγκλε. Äh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει δυστυχώς να πω πως και εγώ πρέπει να φύγω στις 12 γιατί έχω μία αντιπροσωπεία της νεοεκλογής σας κυβέρνησης της Κυργιζίας και βεβαίως είναι αγένεια να αφήσω τους ανθρώπους να περιμένουν στην είσοδο είναι και υψηλό επίπεδο αντιπροσωπεία θα προσπαθήσω λοιπόν και εγώ να κάνω λίγο γρήγορα. Ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να παρουσιάσω την έκθεση αυτή την Επιτροπή πρέπει να δούμε εδώ πέρα ποια ήταν η αιτία αυτής της έκθεσης η Ισπανική Προεδρία το θέμα αυτό της γυναίκες της υπαίθρου ε, το είχε ως μία από τις τρεις προτεραιότητες της και μετά την Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου το ζήτημα αυτό παρά το ότι υπήρχε μία μεγάλη διάσκεψη ε, κάπου χάθηκε αλλά κάποιοι θεωρούσαν πως είναι ένα σημαντικό το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε ειδικά σε σχέση με τη συζήτηση για την κοινή γεωργική πολιτική να αναφερθούμε ειδικά στον δεύτερο πυλώνα και στη, να δοθεί ένα πρόσωπο στις γυναίκες υπαίθρου. Ρώτησα λοιπόν αρκετούς συναδέλφους, ε, έλαβαν το σχέδιο όσοι το ζήτησαν και στις ομάδες, αλλά ε, ήρθα σε επαφή και με ενώσεις αγροτισών, ε, Βεβαίω ξέρετε πως ε, είναι περιορισμένο το μέγεθος μιας έκθεσης που αφορά μόνο τις 6.000 ε, ε, λέξεις ε, θεωρώ λοιπόν πως μπορούμε εδώ πέρα να το συμπληρώσουμε αυτό με τροπολογίες και θα ήθελα να ζητήσω εδώ την βοήθειά σας. Έχει χωριστεί σε πέντε κομμάτια, δύο αφορούν τις αιτιολογικές σκέψεις για τις γυναίκες, για, τους πολυλειτουργικούς, ε, για την πολυλειτουργική ύπεθρο και μετά η ύπεθρος ως ε, χώρος οικονομίας και γυναίκες στη γεωργία. Και να παρουσιάσω κάποια σημαντικά σημεία. Εμείς θεωρούμε και ολόκληρη η Επιτροπή Γεωργίας εδώ πέρα με στηρίζει πως οι γυναίκες είναι η σπονδυλική στήλη της Γεωργίας και της υπαίθρου ολόκληρης η παρουσία τους είναι όλο και πιο έντονη και άρα έχει σημασία να τονίσουμε το ρόλο τους και στις γεωργικές ε, επιχειρήσεις και στην Ήπεθρο παίζουν έναν πολύ λειτουργικό ρόλο και πρέπει βεβαίως να πούμε και ποιες είναι και οι επιδόσεις που έχουν άντρες και γυναίκες χρειάζονται μια προοπτική στην Ήπεθρο. Τι εννοούμε εδώ πέρα, δηλαδή έχουμε Ήπεθρο σε πολλά σημεία από την οποία φεύγουν οι εκπαιδευμένες γυναίκες και αδειάζει και μένει η Ήπεθρος χώρα χωρίς γυναίκες. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα ένα δυναμικό το οποίο εξαφανίζεται και αυτό ανησυχεί πολλά κράτη-μέλη, οπότε είναι κάτι το σημαντικό. Αναρωτιόμαστε ποιε μπορούν να είναι οι ανάγκες αλλά και οι δυνατότητες των γυναικών για να μπορέσουν να ενσωματωθούν καλύτερα Το ένα θέμα είναι η σύνδεση επιχειρη... γυναικών που έχουν επιχειρήσεις ε, και πώς θα συνδεθεί αυτό με την οικογένεια ή πως μια γρότησα γυναίκα, τέλος πάντων μια γυναίκα η οποία είναι ελεύθερη επαγγελματίας να μπορέσει να ζήσει ή όταν είναι αγρότησα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα είτε παιδικών σταθμών είτε φροντίδας των ηλικιωμένων, τι χρειάζεται από πλευράς εκπαίδευσης, κατάρτισης ε, κτλ. Ε, βεβαίως δεν έχουμε κάποια δεδομένα στα οποία να βασιστούμε, γι' αυτό είναι δύσκολο ε, με αυτά τα οποία υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε πάρα πολλά καλά παραδείγματα, αλλά είναι δύσκολο να βρούμε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, να διαπιστώσουμε ποιες είναι και να τις μεταδώσουμε. Οι αγρότησες, και αυτό ήταν θέμα και στην συζήτηση, έχουν βεβαίως ε, τις υποχρεώσεις οι οποίες εννοείται ότι τις αναλαμβάνουν αλλά πρέπει να ανταποκρίνονται και στα δικαιώματα ε, αυτό το οποίο κάνουν. Δηλαδή να εκπροσωπούνται στις ενώσεις αγροτών, να συμμετέχουν στα έσοδα και κοινωνική ασφάλιση. Είναι λοιπόν σαφές και κατέστη σαφές ε, στα διάφορα πως υπάρχει διαφορά στην νομοθεσία, αλλά είμαι παρόλα αυτά πεπισμένη πως πρέπει να το συζητήσουμε. Η διατύπωσή μου, δηλαδή να υπάρχει εκπροσώπηση ε, στις διάφορες ενώσεις λοιπά Μου ζητήθηκε ε, εκεί που μου απάντησαν ε, να υπάρχει ποσόστοση για τις γυναίκες μέχρι και 40%. Θα δούμε τώρα πώς θα περάσει αυτό στις διάφορες αναγνώσεις. Τον Ιούνιο είχαμε ήδη μία πρώτη συζήτηση και το συζητήσαμε ε, μακρόν αυτό το θέμα. 28 Σεπτεμβρίου μετά οργανώσαμε και ένα εργαστήριο και τώρα 26 Οκτωβρίου παρουσίασα την έκθεση αυτή στην Επιτροπή Γεωργίας και Μέχρι τις 16 Νοεμβρίου μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες και 26 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας και το Μάρτιο θα πάμε στην ολομέλεια, Οπότε καιρό έχουμε για να γίνουν συζητήσεις και βεβαίως είμαι ανοιχτή σε αυτό. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Και εγώ σας ευχαριστώ διότι πιστεύω ότι ανταποκριθήκατε ακριβώς αυτά που θέλαμε, μας δώσατε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμασταν. Χρονοδιάγραμμα τώρα, το είπατε και αυτό, είναι σαφέστατο. Μέχρι τις 16 Νοεμβρίου για τις τροπολογίες και στη δική σας επιτροπή ψηφοφορία πολύ αργότερα. Έχουμε χρόνο λοιπόν για να συζητήσουμε τις τροπολογίες στην Επιτροπή Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Και τώρα λίγη συνεδρίαση μας καθεαυτήν και θα μείνουν μόνο οι συντονιστές για τη συνεδρίαση τους. Παρακαλώ όσους δεν είναι συντονίστριες να φύγουν από την αίθουσα γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ.